So, ich bitte doch alle die Plätze einzunehmen. Und äh, Παρακαλώ καθίστε. Ελέγχουμε λίγο την ε, ατμόσφαιρα. Να έχουμε τη σωστή ποιότητα στον αέρα. Σε αυτή την αίθουσα Συχνά το κάνουμε, να ελέγξουμε δηλαδή τον αέρα. Εκτός από τα ιστονικά και τα μαλτέζικα, έχουμε όλες τις άλλες γλώσσες σήμερα. Δεύτερη ανακοίνωση. Έχουμε τριμερείς διαλόγους. Ο πρώτος αφορά τις κλινικές δοκιμές. Εχτες έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος για την έκθεση Μπελιέ Δεύτερος τριμερή διάλογος θα γίνει στι 2 Νοεμβρίου και μετά θα γίνει και ένας τεχνικός τριμερής. Ε, να εγκρίνουμε τα πρακτικά, δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. οπότε προχωράμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Ελπίζω πως όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν φέρει και τις κάρτες ψηφοφορίας τους. και θα τις έχουν ε, βάλει στη, στο μηχάνημα. Μήπως κάποιος έχει ξεχάσει την κάρτα του. Frau Taylor ist jetzt auch versorgt und damit können wir jetzt, können wir jetzt anfangen, über das Verhandlungsmandat abzustimmen. Ωραία. Λοιπόν, τότε μπορούμε να ψηφίσουμε για τη διαπραγματευτική εντολή για το συγκεκριμένο θέμα. δηλαδή άνοιγμα διαπραγματεύσεων για συμφωνία, με στόχο μάλλον, συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση υπό το άρθρο 50 όπου η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συμμετέχει. Ηλεκτρονική θα είναι η ψηφοφορία και όχι η διανατάσταση της χειρός. Χρειαζόμαστε 36 υπέρ. για να υπάρχει απαρτία και να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, η οποία αρχίζει τώρα. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε δύο παραπανήσιους σοσιαλιστές. Τώρα εντάξει. Τέλος ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 18 κατά. Μία αποχή. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε την εντολή για τις διαπραγματεύσει. Οπότε θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Σημείο 5. Αυτή είναι η έκθεσή μου. Μπορούμε να ψηφίσουμε και εδώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία αποχή. Στη συνέχεια πάμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης. Έχουμε τα διοκτώνα. Εδώ θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται ναι 30 και 32 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 31 και 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 και 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι, συγγνώμη, απορρίπτεται διορθώνει ο πρόεδρος, σας επαληθεύσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. 34 και 35 από κοινού ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ Α, έχουν καταπέσει οι δύο επόμενες 36 37 39 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 έχει καταπέσει και περνάμε στην συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 47 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 έχει αποσυρθεί 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20 ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Τρόπολογια 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 και 23 υπέρ. Κα... Α, όχι, έχουν καταπέσει. 24. Ναι, επίσης έχει καταπέσει. Και πάμε στην 25. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 περ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κατά συνέπεια, περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα στο σύνολό του και εδώ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται... Τώρα θα ψηφίσουμε για την εντολή. Ψηφίζουμε. Ψήσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και ευχαριστώ για αυτή την πολύ μεγάλη πειθαρχία που επιδεικνύεται. Συνεχίζουμε. Jetzt geht weiter mit der Abstimmung zur grünen Infrastruktur. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τις πράσινες υποδομές. Είστε όλοι έτοιμοι. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά Ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 20. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ α όχι αυτή είχε καταπέσει 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος. Για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα λοιπόν απορρίφθηκε. 28 υπέρ. Κατά. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Υπέρ της 28. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές α, μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος Απο, απορρίπτεται τι θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για 33 Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Απο... Α, έχει καταπέσει μάλιστα. Όχι, δεν έχει καταπέσει. Την ψηφίζουμε 37 υπέρ. Κα... Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41. Όχι. Απαλήθευση για 39. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα 41 κυρία Ρέμερς είναι η δική σας τροπολογία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 43 όχι 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά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 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62 Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 63 υπέρ κατά Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 έχει καταπέσει. Υπέρ ε, της 67 κατά αποχές δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 67. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 69. 8 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές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 απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί 17. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται ομόφωνα. Συνεχίζουμε. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Θέλω να πω ότι η ποιότητα του αέρα και η θερμοκρασία στην αίθουσα, δεν ξέρω αν είναι δοκιμή ή όχι, πάντως... Δουλέψαμε υπό δοκιμαστικές συνθήκες και περνάμε τώρα ε, στην έκθεση της Julie Gerling για το μέλι. Θα περιμένω λίγο. Όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Και μετά θέλω ησυχία στην αίθουσα, ώστε η Julie Gerling να μπορέσει να πάρει τον λόγο. Vielleicht können sich Mitarbeiter mit ihren Chefs. Σας παρακαλώ. Όσοι θέλετε να μιλήσετε από τους υπαλλήλους με τους ανωτέρους σας, παρακαλώ εκτός εθούσης. Η Τζούλη Γκάλινγκ πάντω θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάρει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ε, μια στιγμή, μια στιγμή. Περιμένετε γιατί πίσω από εσά γίνεται μια συζήτηση και δεν θέλω να σας δυσκολεύει. Παρακαλώ, τώρα έχετε το λόγο. Οι περισσότεροι από όσους έχουν ασχοληθεί με την έκθεση αυτή γνωρίζουν το υπόβαθρο. 19 Δεκεμβρίου πέρυσι ξεκίνησε η έκθεση. Πραγματικά είναι από τα θέματα τα οποία έχουν παραμείνει εκτός ψηφοφορίας ε, περισσότερο. Θα συνοψίσω λιγάκι περί τίνος πρόκειται. 2011 είπαμε για τα στατικά του μελιού. Για την γύρι και υπήρξε περίπτωση στο δικαστήριο και είπαμε ότι θα πρέπει να αναφέρεται σαν συστατικό. Πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση της γενετικά τροποποιημένης ε, γύρισης, εφόσον είναι πάνω από 9%. Τώρα έχουν, έχει υπάρξει σύγχυση βέβαια με τους παραγωγούς που δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να βάζουν στις ετικέτες για τις εξαγωγές, τις συμφωνίες που κάνουν για τις εξαγωγές και τα Είναι Συνεπώς, η Επιτροπή έκανε μία πρόταση προσπαθώντας να επαναφέρει τα πράγματα στα πριν της ε, απόφασης του δικαστικού δικαστηρίου να το θεωρήσει σαν ένα φυσικό συστατικό του μελιού. Εγώ έχω συναντηθεί με αρκετού ε, μελισσοκόμους και με καταναλωτές που θεωρούν ότι είναι ένα φυσικό προϊόν το μέλι. Εγώ στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής, η οποία λέει ότι αποτελεί μέρος του μελιού. Δεν προστίθεται από τους μελισσοκόμους, οι μέλισσες προσθέτουν το συστατικό αυτό, οπότε συμπεριλαμβάνεται στα φυσικά συστατικά. θα ήταν παρατυπία εάν υπάρξει κάτι διαφορετικό στην αγορά. Πάντως η απόφαση λέει ότι χρησιμοποιούν το θέμα αυτό σε θέλουν να ενισχύσουν τη συζήτηση για τα γενετικά τροποποιημένα. Τι γίνεται λοιπόν όταν είναι πάνω από 9% για οποιοδήποτε συστατικό. Εάν λοιπόν τη γύρη την υπολογίζουμε σαν ε, ποσοστό, έτσι κι ποτέ δεν θα ξεπερνάει το όριο. Αν όμως το θεωρήσουμε σαν συστατικό, τότε πρέπει να δούμε το ποσοστό της γύρης. Και θεωρητικά αυτό σημαίνει ότι η γενετικά τροποποιημένη γύρης, η οποία θα υπολογίζεται σαν ποσοστό της συνολικής γύρης, θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα. Πρέπει να τη θεωρήσουμε δηλαδή συστατικό για να υπάρχει και πάνω στην ετικέτα. Και αυτό λοιπόν και εγώ συστήνω το εξή στην εκθεσή μου. Το όριο το 0,9% έχει να κάνει με όλα τα τρόφιμα. Αν εδώ κάνουμε μια εξαίρεση με το μέλι, τότε θα επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τους εξαγωγείς και τους μελισσοκόμους, γιατί θα πρέπει να περνάνε από εξετάσεις τα προϊόντα τους. και πώς θα εφαρμόσουμε ένα τέτοιο μέτρο. Ακόμα δεν έχουμε επαρκείς ε, μεθόδους μέτρησης για το ποσοστό της γενετικά τροποποιημένης γύρης μέσα στην υπόλοιπη γύρη. Οπότε πώς θα είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο ξεπερνιέται ή όχι το 0,9%. Εγώ αντιλαμβάνομαι βέβαια τα κίνητρα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές Υπάρχουν θεμητές ανησυχίες για την συνύπαρξη αυτή και για το ότι πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες κάθε φορά που υπάρχει γενετικά τροποποιημένο προϊόν. Όμως, τότε πρέπει να δούμε τον ε, κανονισμό για τα γενετικά τροποποιημένα και τις ετικέτες και όχι την οδηγία για το μέλι. Κινδυνεύει λοιπόν ο τομέας του μελιού από αυτήν τη συζήτηση και πρέπει πιστεύω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς θα συνεχίσουμε. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα να δείτε την μεγαλύτερη εικόνα και αν θεωρήσουμε συστατικό τη γύρι, τότε ε, μάλλον ε, οδηγούμε σε λάθος δρόμο τους καταναλωτές και πλήττουμε και τους μελισσοκόμους και μελισσοπαραγωγούς, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θέλουμε να είναι η πρόθεσή μας. Ευχαριστούμε. Ο... Παρακαλώ, ο κύριος Πέτελε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συστηθώ πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε. Γιατί εκτός από Ευρωβουλευτής είμαι και μελισσοκόμος. Δεν είμαι πολύ μεγάλος μελισσοπαραγωγός, δεν έχω να κάνω με άλλες υπήρους. Είμαι επίσης και καταναλωτής και έτσι και πελάτης. Οπότε μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να ξέρουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για τη συζήτησή μας και το βγά ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο θα κερδίσει το συστατικό η περιεκτικότητα. Εγώ νομίζω ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πάνω απ' όλα για το κατά πόσο το μέλι το οποίο αγοράζουν έχει γενετικά τροποποιημένη γύρι ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ευαισθησία και μεγαλύτερη πόλωση μάλιστα σε αυτά τα θέματα. Εγώ δεν θα ήθελα εμείς εδώ να διχαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρίτο δρόμο εδώ. Που να προσανατολίσετε περισσότερο στα συμφέροντα του καταναλωτή. Αλλά και στην αγορά. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εδώ για την περίπλοκη τεχνολογία που ισχύει όσον αφορά τις ποσότητες, τα ποσοστά κλπ. Με τις τροπολογίες μου προτείνω να ακολουθήσουμε το δικαστήριο και να τη θεωρήσουμε συστατικό την γύρη του μελιού. Ξέροντας όμως τα προβλήματα που αναφέρθηκαν κιόλα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με μια απλή λύση. Το μέλι, η μέρος του μελιού θα έχει ετικέτα ως ε, ε, μέλι το οποίο έχει γενετικά ε, τροποποιημένη γύρι ή στο οποίο έχουν βρεθεί ίχνη γενετικά τροποποιημένης γύρης. Όποιος θέλει σε θελοντική βάση μπορεί να δώσει το μέλι του, να περάσει από τα τεστ και έτσι να πάρει την ετικέτα μελιού που δεν έχει γενετικά τροποποιημένη γύρι. Με αυτόν τον τρόπο σε κεντρικό σημείο θα βάλουμε την επιλογή του καταναλωτή και η ποιότητα επίσης θα έχει αντίκτυπο στις τιμές. Οι μελισσοκόμοι λοιπόν οι οποίοι θέλουν και θα μπορέσουν να πείσουν τους καταναλωτές θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις μάρκες και τις ετικέτες που λένε ότι έχει περάσει τα τεστ το μέλι τους και δεν βρέθηκαν ίχνη γενετικά τροποποιημένης γύρης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στην Κομισιόν και το Δικαστήριο. Δύσκολο είναι να αποφασίσουμε κατά πόσο είναι στοιχείο της σύνθεσης συστατικό. Η αγορά νομίζω θα αποφασίσει πιο εύκολα με τη λύση που σας πρότεινα. Αυτό προτείνω. Για να αποφύγουμε την πόλωση και παρετέρω συζήτηση για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ευχαριστούμε. Äh, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την Τζούλη Γκέρλινγκ καταρχήν αλλά εάν αρχίσουμε να λέμε ότι η γύρι είναι συστατικό, τότε ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Γνωρίζω ως παραγωγός ότι το μέλι είναι ένα καθαρό προϊόν που παράγεται από τις μέλισσες γιατί αν μιλάμε για τη γύρι όχι ως συστατικό, αλλά ως ε, πρόσθετο, τότε πάμε, ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή για το γάλα μπορούμε να πούμε σε αντίστοιχη περίπτωση λακτόζη, τι θεωρείται, είναι συστατικό ή προσθετικό. Ε, το ίδιο αφορά και σε άλλους, και άλλους τομείς, ε, δηλαδή ας πούμε στο αυγό, ο κρόκος τι είναι, συστατικό ή όχι. Τι είναι το ασπράδι, τι είναι ο κρόκος. Για μας το ζήτημα είναι απόλυτα σαφές. Το αυγό ε, είναι ένα πλήρες ε, προϊόν το οποίο έχει συστατικά. Τα συστατικά αυτά είναι το ασπράδι και ο κρόκος. Και σε αντίστοιχη περίπτωση η μέλισσα παράγει μέλι και την γύρι εμέσως. Άρα μιλάμε για αναπόσπαστο συστατικό του μελιού. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ε, λέξεις. Είναι εντελώς λανθασμένος αυτός ο διαχωρισμός. Στην περίπτωση της γύρης, τι μιλάμε, για τι πράγμα μιλάμε, για συστατικό ή όχι, πρόκειται για γενετικός τροποποιημένο οργανισμό ή όχι. Ε, θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστο συστατικό του μελιού. Και υπ' αυτή την έννοια έχω υποβάλει τροπολογίες. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το Κοινοβούλιο επιμένει. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ακόμα και στα παραρτήματα, ίσως η Επιτροπή μπορεί να δράσει πιο αποτελεσματικά, αλλά θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να κάνουμε εμείς υπερβάσεις. Εάν λέμε λοιπόν ότι είναι συστατικό και όχι στοιχείο της σύνθεσης, τότε αυτό θα πρέπει να ισχύσει για σωρία προϊόντων και ανοίγουμε το κουτί της παντόρας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι το θέμα της κότας και του αυγού σε αυτή την περίπτωση. Ε, σε σχέση με τους ε, τρυποποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορεί να οδηγήσει και στην απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι οι μέλισσες ε, διαδίδουν αυτή την γενετικό, τροποποιημένη γύρι. Πρόκειται για επικίνδυνο προϊόν. Θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα ανιχνευσιμότητας, άρα θα πρέπει να πιάσουμε τη κάθε μέλισσα και να υπάρχει σήμανση σε κάθε μέλισσα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανιχνεύσης. Επίσης χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης των μελισσών. Δεν γνώριζαν αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσει του σύγχρονου καταναλωτή. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε DVD ή ηλεκτρονικά μέσα ανείχνευσης. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικές προβολές προς τις μέλισσες, να γίνει ένα brainstorm για να ξέρουν τι συμβαίνει. Ε, σε αυτή την περίπτωση ίσως υπάρξει επιμόλυνση από την χρήση αυτή της συγγύρισης. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η ειδική κατάρτιση των ε, μελισσών, οι οποίες να απομακρύνουν αυτή τη γύρη πριν πάει στο μέλι. Εδώ πρόκειται για μία νομική πρόκληση όταν πρόκειται για τέτοιες ε, δράσεις και ίσως οι εκπρόσωποι των μελισσών στα δικαστήρια μας πούν ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι η γύρη αυτή είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος Και έτσι σε αυτή την περίπτωση οι κίνδυνοι που απορρέουν από το μέλι είναι πολύ πιο μακρινή από, έναν, ε, από ένα αστεροειδές το οποίο θα μπορούσε να μας πλήξει ανα πάσα στιγμή. Πολύ γελία πράγματα πολλές φορές και νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση της Τζούλη. Είναι η μόνη λογική μας πράξη. Ευχαριστούμε. Η Πιλάρα Ευχαριστώ. Χωρίς να είμαι ηρωνική όπως ο κύριος Ντέιβις, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, πρόταση Γκέρλινγκ και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για στοιχείο της σύνθεσης και όχι συστατικό. Μιλάμε για ένα 0,9% άρα είναι παράλογο να μιλήσουμε για ε, σήμανση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ας πούμε ο αραβόσιτος δεν ε, χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση Γκέρλινγκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια μελισσοκόμων. Συμφωνώ με τον Chris Ντέιβις και με άλλους ομιλητές Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ορμηνεύσουμε τις μέλισσες για το πώς θα πρέπει να δράσουν μπορούν ε, να υπερίπτανται όπου θέλουν. Και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί στην ακτίνα τους. Γι' αυτό υποστηρίζω την Julie Gerling. Αυτά είναι τα δεδομένα και δεν χρειάζεται να τους δίνουμε ε, άλλες διαστάσεις στα πράγματα από αυτές που έχουν. Κλείνοντας θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Ήδη αναφέρθηκαν τα περισσότερα επιχειρήματα που θα ήθελα να προβάλλω. Πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τα σοβαρότερα συμφέροντα του τομέα της μελισσοκομείας όπως ορίζει και η μελέτη αντικτύπου γιατί θεωρούμε ότι το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν που ε, εκμεταλλεύονται οι μελισσοκόμοι. Η γύρι αποτελεί στοιχείο της σύνθεσης και όχι συστατικό. Και αυτό δεν είναι επινόηση κανενός. Πρόκειται για ένα στοιχείο της σύνθεσης που παράγεται φυσικά. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την απόφαση του δικαστηρίου λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ε, ε, με βάση τον κανονισμό 1829 κάθετος 2003. Θεωρούμε ότι πρόκειται για παραγωγή συστατικού τροφίμων χωρίς ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και θα πρέπει να υπάρχει ε, σήμανση όπου θα πρέπει να γίνεται και σε άλλη περίπτωση τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα 0,9%. Ε, Αυτό είναι το όριο επισήμανσης έτσι κι αλλιώς που ισχύει. Άρα δεν πρέπει να συγχαίουμε αυτή τη συζήτηση ως προς την συνύπαρξη που ε, αφορά μια άλλη συζήτηση που δεν σχετίζεται με το μέλη. Θεωρούμε λοιπόν μετά τις συζητήσεις, τις σημερινές, ότι ότι υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Τέλος, η εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τα μέλη που υποστηρίζουν την έκθεση. Προβάλλεται μία ε, νέα ιδέα από από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δοκιμές γύρω από την ύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και πώς ορίζονται στη σήμανση. Νομίζω λοιπόν ότι από τεχνικής πλευράς θα ήταν πολύ δύσκολο να ενσωματωθεί κάτι τέτοιο, αλλά θα το σκεφτώ εκτός συνεδρίασης πριν ψηφίσουμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι μέσα στα πλαίσια συμβιβασμών. Είναι δύσκολος αυτός ο συμβασμός γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο συμφωνούμε ή όχι. Δηλαδή θεωρούμε, θεωρούμε ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύνθεσης ή συστατικό. Ως προς τα άλλα ε, θέματα που εφήγησαν, όλοι δεχόμαστε ότι εδώ δεν πρόκειται για θέμα συνύπαρξης ούτε σήμανσης με βάση τους ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Γιατί μας χρειάστηκαν δέκα μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το ε, συμπέρασμα, διότι έγιναν ζωηρές ε, συζητήσεις στην αρχή και δεν ακούσαμε αυτά τα ζωηρά επιχειρήματα σήμερα και επειδή και εμείς ε, ε, εκπονήσαμε μία μελέτη αντικτύπου, είδαμε ότι επιλύθηκαν τα προβλήματα και δεν υπάρχουν πλέον οι ανησυχίες που είχαν ε, αρχικά εκφραστεί. Αυτή είναι η θετική έκβαση των πραγμάτων. Σας και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκέρλιν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Η Άγκρη θα ψηφίσει στις 5 Νοεμβρίου και στην Έμβη θα ψηφίσουμε στις 27 Νοεμβρίου. Και ακόμα δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία για την συζήτηση στην Ολομέλη. Ως προς την έκθεση Τελάνγκε δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πρόκληση να εξετάσω αυτό το θέμα μετά μάλιστα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Έτσι καλώς είμαστε περιορισμένοι για την έκταση της ε, έκθεσης πρωτοβουλίας. Θα μπορούσα να είχα γράψει δύο και τρία φορές παραπάνω. Και αυτό προσπάθησα να περιοριστώ στο κύριο κομμάτι, στην ουσία του θέματος. Είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας ακριβώς επειδή είχαν υπάρξει διάφορες απάτες στον τομέα των τροφίμων τον τελευταίο καιρό. Το κρέας αλόγου είναι το τελευταίο, αλλά πριν από αυτό είχαμε και διάφορες χωστικές ουσίες στις καραμέλες, είχαμε ε, αλάτι το οποίο κανονικά δεν είναι για κατανάλωση από τον άνθρωπο που βρέθηκε στο ψωμί κλπ. Τώρα, έχουμε περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις τελευταία. Υπάρχει ένα παράδοξο. Από τη μια μεριά, τα τρόφιμα στην Ευρώπη ποτέ δεν ήταν τόσο ασφαλή. Ως Ευρωπαίοι δηλαδή έχουμε 260 φορές παραπάνω πιθανότητες να πεθάνουμε από γρήπη από ότι από κάποιο τρόφιμο που καταναλώνουμε. Είναι δηλαδή ασφαλή τα τρόφιμά μας. Από την άλλη μεριά όμως, ακριβώς επειδή πρόσφατα είχαμε διάφορα σκάνδαλα, οι καταναλωτέ το 1 τρίτο των καταναλωτών τουλάχιστον, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στι ετικέτε που βλέπουν στα προϊόντα. Τι είναι η απάτη λοιπόν. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, Πολιτείες, εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε αποφασίσει για ένα συγκεκριμένο ορισμό. Δηλαδή δεν ξέρουμε τελικά τι είναι ακριβώς αυτό το φαινόμενο που θέλουμε να εξετάσουμε. Φυσικά και υπάρχει νομοθεσία όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων. Έχουμε επίσης στο, στη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα ότι δεν πρέπει οι ετικέτες να οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα των καταναλωτή. Έχουμε ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων, αλλά τελικά οι απάτες αυτές τελικά πώς ξεφεύγουν από τους ελέγχους. Σίγουρα εμείς αυτό που έχουμε δει είναι την κορυφή του παγόβουνου. Το ξέρουμε αυτό. Όμως, τι υπάρχει πιο κάτω στα πιο κάτω στρώματα αυτά είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα ξέρουμε καλά. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε για έναν ορισμό στην Ευρώπη, για το τι είναι αυτό το φαινόμενο. Τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο μηχανό, για παράδειγμα, η μη συμμόρφωση με την ομοθεσία για τα τρόφιμα, η παραπλάνηση των καταναλωτών. Ω δεύτερον, το ότι γίνεται σκόπιμα η απάτη αυτή γιατί εντάξει κατά λάθο μπορεί πάντα να συμβεί κάτι εδώ, πρέπει να υπάρχει και αυτό το στοιχείο το ότι είναι σκόπιμο. Και το τρίτο, ότι γίνεται για λόγους οικονομικού κέρδου. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα στοιχεία όμως, δεδομένα. Ορισμένες χώρε μέλη κάτι έχουν, άλλες χώρε μέλη όμως δεν έχουν σχεδόν τίποτα. Συνεπώ πρέπει να φροντίσουμε να συγκεντρώσουμε δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα για το φαινόμενο. Τώρα οι κατηγορίες ε, των απατών που έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα θυμόσαστε ότι υπήρχε και ένα θέμα με το χυμό ροδιού και εκεί που είχε ανακατευτεί με πορτοκάλι. Έχουμε επίσης το κρέας, με το κρέας αλόγου πρόσφατα. Ε, προϊόντα που δεν είναι βιολογικά και τα οποία πολλούνται ως βιολογικά. Πράγματα τα οποία ε, βέβαια παραπλανούν τον καταναλωτή. Επίσης υπάρχει η απομίμηση προϊόντων. Νομίζει κανείς ότι αγοράζει ένα εγκυμένα περιφερειακό προϊόν, ενώ τελικά δεν είναι τέτοιο. Προϊόντα επίσης τα οποία ακούγονται πολύ και αναφέρονται πολύ στην ε, νομοθεσία. Είναι το ελαιόλαδο, τα ψάρια, τα βιολογικά τρόφιμα, αλλά και το μέλι πριν αναφερθήκαμε στο μέλι και το σιρόπι σφενδάμου. Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε. Ο κίνδυνος απάτης πάντως είναι υψηλότερος όταν ο κίνδυνος εντοπισμού είναι περιορισμένος και το οικονομικό κέρδος είναι μεγάλο. Στην Ευρώπη λοιπόν ο εντοπισμός δυστυχώς δεν είναι αρκετός προς το παρόν. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την ασφάλεια τροφίμων χωρίς να σκεφτόμαστε το θέμα της παραποίησης, της αλλίωσης όπως λέγαμε πριν. Σίγουρα είναι περίπλοκη η αλυσίδα η διατροφική. Το να υπάρχει εμπόριο Πολύ ωραία. Πάντω η αλυσίδα αυτή διατροφική είναι πολύ πιο περίπλοκη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Έπειτα διασυνοριακά κυκλοφορούν τα τρόφιμα και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται συνεργασία Λοιπόν, η Europol, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσουν, γιατί αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη είναι περιορισμένα. Και στο κάτω-κάτω το ένα κράτος μέλος διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ πιο ανοιχτό στο να κάνει ελέγχου και να προσπαθήσει να εντοπίσει τέτοιες απάτες από ότι άλλες χώρες μέλη. Για παράδειγμα, η δικιά μου η χώρα δεν ήταν πολύ διατεθειμένοι να συνεργαστεί με την Κομισιόν ή με την Europol για να εντοπιστούν, ε, όπως έγινε με το κρέας για παράδειγμα, δεν συνεργάστηκαν πολύ. Συνεπώς, οι έμποροι τροφίμων πρέπει να συνεργάζονται, να δέχονται τους ελέγχους. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες και διαρθρωτικές αδυναμίες στο σύστημα παραγωγής τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρόφιμα, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν ήταν τόσο ασφαλή όσο σήμερα. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σύνορα, ότι υπάρχει εθνική κυριαρχία και η εθνική αρμοδιότητα ο έλεγχος των τροφίμων, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να εντοπίζονται δύσκολα οι παρατυπίες. Το είδαμε και με το κρέας αλόγου. Πόσο δύσκολο ήταν να εντοπίσουμε ε, το πρόβλημα επειδή το πριόν είχε εγκαταλείψει τη χώρα. Τελικά είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αρχή η οποία είναι αρμόδια να εντοπίσει, να κυνηγήσει, να διώξει τους υπεύθυνους. Ενημερώθηκαν οι Βρετανικές αρχές, η Ολλανδία, η Europol, αλλά τις πληροφορίες αυτές οι οποίες κυκλοφόρησαν σίγουρα δεν τις χειριστήκαμε αρκετά γρήγορα και αρκετά καλά. Εγώ κάνω κάποιες προτάσεις, σε θεσμικό πλαίσιο δηλαδή τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Πέρα από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία ομάδα για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, είναι βέβαια στην αρχή. Θα ήταν καλό λοιπόν να δούμε και τον ρόλο της υπηρεσίας που έχουμε στο Δουβλίνο για τα τρόφιμα. Να τον ενισχύσουμε, αλλά να γίνει ίσως και πιο πολιτικός. Οι εκθέσεις που εκπονεί ο οργανισμός αυτός μερικές φορές είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν δίνουμε ιδιαίτερη συνέχεια. Πάλι με το κρέας αλόγου υπήρξε στην έκθεση του γραφείου τα διάφορα στοιχεία. Η γνώση υπήρχε δηλαδή. Πόσο εύκολο δηλαδή είναι να καταλήξει κανείς σε απάτες με το κρέας αλόγου. Τι κάναμε με την έκθεση αυτή, τίποτα. Η συζήτηση με την υπηρεσία αυτή, με τον οργανισμό αυτών λοιπόν πρέπει να γίνεται πιο πολιτικά ετησίως εδώ. Να ρωτάμε ποιοι είναι οι στόχοι σας για τον επόμενο χρόνο κτλ. Να έρχονται εδώ και να τα ακούμε όλα αυτά. Όσον αφορά την νομοθεσία τώρα. η νομοθεσία πρέπει να θεωρηθεί όσον αφορά τους ελέγχους που κάνουν οι χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πολύ διακριτικό βήμα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάει πιο μακριά. Με το παράδειγμα πάντα της απάτης με το κρέας αλόγου σε ένα συγκεκριμένο χώρο, 30.000 ευρώ είναι το πρόστιμο. Ενώ 65.000 ευρώ κερδίζει κανείς από ένα κοντέινερ με την απάτη αυτή. Άρα οι κυρώσεις δεν είναι αρκετά αυστηρές. Έπειτα κάνω και μια πρόταση για το business to business ετικέτες. Δηλαδή να γίνουν πιο αυστηροί κανόνες και πιο επαγγελματική η επίθεση αυτή ετικετών. Και σίγουρα δεν μπορούμε από μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι ένα θέμα και κοινωνικής ευθύνης. Για παράδειγμα, όταν είσαι έμπορος και πουλάς τρόφιμα να σε νοιάζει το από πού προέρχονται τα συστατικά των τροφίμων σου. Να μπορείς και εσύ να δώσεις κάποια εγγύηση. Πολλές ε, επιχειρήσεις το προσέχουν αυτό. Υπάρχουν πολλές εθνικές και διεθνείς τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, οι ελεγκτικές αρχές. Φαίνεται ότι οι φορείς ελέγχου δουλεύουν όπως η αστυνομία περίπου. Στη Δανία για παράδειγμα ή στην Ιταλία έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες στον εντοπισμό διατροφικών απατών. Πολλοί από τους ελέγχους όμως είναι γνωστοί από πριν Έτσι προσπαθούν και εντοπίζουν εκ των προτέρων από πού μπορεί να προέρθει ο κίνδυνος. Αυτά προς το παρόν. Αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία που έχω συμπεριλάβει στην έκθεση αυτή. Τώρα περιμένω τα σχόλια των συναδέρφων και είμαι διατεθειμένη τροπολογίες να ετοιμάσουμε από κοινού μαζί γιατί σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί κανείς να πει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Ζήλ Πονιών. Σκιώδη συγητής. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε έναν τόνο αλλαντικών και δύο τόνους ε, ψαριών ή ψαρικών που στην ουσία ε, μπορούν να οδηγήσουν σε ε, τροφική δηλητηρίαση. Αυτό αφορά και είδη ζαχαροπλαστικής και αυτό το βλέπουμε σε 29 χώρες όπως δείχνει η Europol. Αυτό δείχνει το μέγεθος ενός φαινομένου το οποίο αφορά την ε, απάτη στο τομέα των τροφίμων. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει να τονίσουμε και την ανάγκη να νομοθετήσουμε σε αυτό το τομέα, διότι όταν μιλάμε για παραχάραξη Μέχρι τώρα μιλούσαμε για ηλική παραχάρηση, δηλαδή ε, σε σχέση με διαφυγόντα κέρδη, πνευματικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Τώρα μιλάμε για παραχάραξη στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής, όπου μιλάμε για πάτες όπου διατρέχει κανείς κινδύνου στην υγεία και την υγιεινή. Πρόκειται για προϊόντα που μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα, τα, τα αγοράζει καλοπροαίρετα ο καταναλωτής, ενώ υπάρχουν θέματα υγείας, υγιεινής καθώς και ασφάλειας. Άρα ε, μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Αυτό απορρέει από τη μελέτη του 2003 για το αλογίσιο κρέας. Στην ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε ρόλο πυροσβέστη και τίποτα άλλο κάτι το οποίο απέχει πόρο από τις ανάγκες μας, θα πρέπει να δράσουμε ανάντι και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, αν και πολλές χώρες δεν συμφωνούν. Θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη νομοθετική δράση, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε βιώσιμα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όπως και η κυρία Αντελάγκε. Συμφωνώ και εγώ θα πρέπει να έχουμε έναν εναρμονισμένο ορισμό της ε, απάτης στον τομέα της διατροφής και των τροφίμων. Όπως και εσείς, όπως και εκείνοι, θεωρώ ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για την μαφία αυτή που δρά στον τομέα διατροφής που απέχει από τον παραδοσιακό τομέα ε, μαφιόζικων δραστηριοτήτων όπως τα ναρκωτικά. Η Γαλλία στους επόμενους μήνες θα ορίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα είναι αναλογικό σε σχέση με τα υπερβολικά κέρδη. Θα υπερψηφίσω την έκθεση, αλλά θα ήθελα να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν ως προς την πληροφόρηση των καταναλωτών, που κάτι το οποίο δεν θίγεται στην πρόταση ψηφίσματος. Βασικός μας στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο κατά των απατών ε, ανάντι. Και θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τη διατροφή, κατά της απάτης δηλαδή, για να καλύψουμε τα χάσματα που υπάρχουν μετά την κρίση στο αλογίσιο κρέας. Επίσης να επεκταθεί ε, η μνήα της προέλευσης του κρέατος από τα στα προπαρασκευασμένα πιάτα. Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει αυτή η υποχρέωση μέσα στα πλαίσια της πληροφόρησης του καταναλωτή για τα παρασκευάσματα αυτά και τα τρόφιμα που ε, έχει οριστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτές οι τροπολογίες θα υποβάλω μέχρι 28 Οκτωβρίου. Επόμενος ομιλητής. Η, επόμενη ομιλήτρια είναι η Κορίντε Λεπάζ. Sorry. Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια, καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή έκθεση και να σας πω ότι υποστηρίζω αυτή την έκθεση υποβάλλοντας και συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία των παραγωγών, των κτηνιάτρων και εκείνων που ασχολούνται με την καταστολή της απάτης στη διατροφική αλυσίδα. Μιλάτε για το πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι ύψης της σημασίας, αν και είναι δύσκολο να εναρμονίσουμε τις κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως θέλουμε να γίνει πρόοδος. Επίσης μιλάτε για τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ε, διατροφική κρίση και την απάτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον τομέα στο σύνολό του, όπως είπε και ο κύριος ε, Παρνιό δηλαδή ανάντι, και να δούμε πώς έχει η ΚΟΑ. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον τομέα της υγείας υγιεινής και περιβάλλοντος. Η απάτη εντάσσεται στον οικονομικό ιστό και οφείλεται και στο κοινωνικό ντάμπινγκ το οποίο διαπιστώνουμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο εκεί. Τρίτον, υπάρχουν ε, οι παράγοντες θέσεις εμπορία όπου δεν υπάρχει σωστή σήμανση η οποία θα έπρεπε να ισχύει σε επίπεδο ε, εκμετάλλευσης παραγωγής αλλά και μεταποιημένων πιάτων. Δηλαδή και εκεί να υπάρχει σήμανση. Χρειάζεται πλήρη σήμανση όλων των κρεάτων είτε είναι βοηδή, χειροειδοί εγωειδή πουλερικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα συστατικά στα μεταποιημένα προϊόντα. Μετά τις εκθέσεις του, των ΜΚΟ στην Ευρώπη και της ΕΠΑ σε σχέση με τις απάτες στη σήμανση στα ψάρια χρειαζόμαστε πλήρη σήμανση σε όλα τα μεταποιημένα προϊόντα. Λυπάμαι διότι η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη και τα φυτικά προϊόντα και ιδιαίτερα τη χρήση φυτοφαρμάκων. Η ευκαιρία κόλλη στη Γερμανία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς και το σκάνδαλο στο Αμερικανικό σιτάρι. Ε, πιστεύω ότι αν υπάρχουν ε, παναλαμβανόμενες απάτες θα πρέπει να απομακρύνονται τα προϊόντα από την αγορά. Κανένα εισαγόμενο προϊόν δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό εάν δεν την χάνει πλήρους ανιχνευσιμότητας από τρίτη χώρα. Θα πρέπει να γενικευθεί το αρνητικό screening για προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Τέλος, σε σχέση με τους ελεγκτές, κυρία Ντελάγκ, θα πρέπει να βασιστούμε στην πείρα μας και να υπάρχουν και τυχαίοι έλεγχοι και δείγματα. Όμως δεν ξέρω κατά πόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να προβούν σε ποιοτικούς ελέγχους τη στιγμή που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα γιατί δεν διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό. Όπως είχαμε πει και σε μία έκθεση το 2002, δεν υπάρχουν αρκετοί κτηνίατροι. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ε, αυξήσουμε την ποιότητα των προϊόντων και όχι να περιστέλουμε το κόστος. Έχουμε τρεις ε, τεχνικούς που ασχολούνται με το θέμα έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτή την αίθουσα. Ελέγχουν τα νέα φίλτρα. Γι' αυτό νομίζω ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς ή καλύτερα από πριν μετά την ψηφοφορία όλα αυτά. Η Τζούλι Γκέρλινγκ έχει το λόγο, συζηγητρία. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή. Γιατί στην εισηγήτρια, με συγχωρείτε, γιατί είναι πολύ επί της η έκθεση της. Δεν νομίζω, δεν βρήκα τίποτα που να διαφωνώ. Θέλω κάποια πράγματα να προσθέσω. Αναγνωρίζω βέβαια τον περιορισμό των ε, λέξεων φαντάζομαι πως όσα θα πω δεν θα την εντυπωσιάσουν την εισηγήτρια, αλλά απλώς ε, για να της δώσω μια ιδέα του τι τροπολογίες θα υποβάλω. Φυσικά και είναι επίκαιρο το ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και ταυτόχρονα εξετάζουμε τις αλλαγές στους επίσημους ελέγχους. Και έτσι έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε κατά τη διάρκεια αυτής τη πρωτοβουλίας και να τα βάλουμε χωριστά σε μια άλλη νομοθεσία. Ο χρονισμός λοιπόν ήταν εξαιρετικός. Τι νομίζω πως μπορούμε να προσθέσουμε. Νομίζω πως μπορούμε όντως να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα του ορισμού των τροφίμων Κομισιόν έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να βρει τους ορισμούς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αναφορά όσον αφορά την απάτη στα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες από κάποια εργαστήρια που κάνουν ε, ελέγχους αυθεντικότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτιαχτούν στάνταρς, προδιαγραφές. Όταν έγινε μια πολύ αποτελεσματική ε, νομίζω εγώ και κέρια επέμβαση μετά από το σκάνδαλο του ε, κρέατος αλόγων όπου γίνανε έλεγχοι σε πάρα πολλές χώρες. Τα, έπρεπε τότε να θεσπιστούν σε ad hoc βάση τα επίπεδα ε, ε, περιεκτικότητας. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο πούμε είπαμε 1%, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν ε, αντικειμενικό ή όχι. Πάντως δεν υπήρχαν επίπεδα, δεν υπήρχαν δηλαδή ανώτατα, κατώτατα όρια κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ε, προδιαγραφές ε, όπως ε, και τα επίπεδα υποκατάστασης, τα επίπεδα μόλυνσης, τι επίπεδα ανοχή θέλουμε, όχι μόνο ποια ποσοστά ελέγχουμε, αλλά και ποιο επίπεδο, για ποιο επίπεδο ελέγχουμε. Πληροφορίες δηλαδή που θα πρέπει να μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιεί μόνιμα, να είναι διαθέσιμες μόνιμα. Και έπειτα οι υπηρεσίες της, FVO, δηλαδή της υπηρεσίας για τα τρόφιμα και τα ζώα, δεν είναι εκπαιδευμένοι ειδικά. Και θα ήθελα να προτείνω αυτό που φαντάζομαι δεν θα ψηφιστεί την Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, επειδή συνδέεται με το, πολυ... με το PDP, αλλά έχουμε και το ορίζοντα 2020 που έχει ένα βασικό πυλώνα για την... τα τρόφιμα και μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε ότι η απάτες στα τρόφιμα είναι ένα βασικό θέμα ε, της, ε, του μείγματος για την ασφάλεια στα τρόφιμα και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν κάποια αυτά τα χρήματα ε, του Horizon 2020 στην ασφάλεια των τροφίμων. Και να, για να αντιμετωπιστούν και οι απάτες στα τρόφιμα. Αυτά θα μπορούσαμε να κάνουμε, να δούμε δηλαδή τι, ποια έρευνα μπορεί να γίνει ώστε τα επίπεδα που ανέφερα να οριστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί βέβαια και η συγκέντρια αναγνώρισε ότι υπάρχουν δημοσιονομικά θέματα. Και έτσι θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Ε, και κάτι τελευταίο, καλωσορίζω τα όσα είπε η συγκέντρια για την ειδική ιδιαίτερη ευθύνη των λιανοπολιτών ήταν εντυπωσιακό να δούμε πόσο άνθησε η δραστηριότητα σε σχέση με την προστασία των, της, των λιανοπολιτών να προστατεύσουν τα σήματά τους. Εμείς θέλουμε να γίνει αυτό. Θα έχουμε μάλιστα επιτάπητος μέσω της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ μία, έναν θελοντικό κώδικα για τους λιανοπολιτές, κυρίως αφορά το κόστος, την κερδοφορία και τις πρακτικές τους. Ε, και το, τις πρακτικές των προμηθευτών και θα ήταν ε, πιθανόν και εύκολο να βάλουμε και τα θέματα της ε, απάτης στα τρόφιμα. Και έτσι θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε πιο γρήγορα θεσπίζοντας στάνταρ και κοινέ προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούζο παρακαλώ. Άλλος, Αλλά προηγουμένως, άλλος ομιλητής. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια για τις προτάσεις της. όντως αναφέρεται το, η απάτη με το κρέας αλόγου. Το θέμα της ασφάλειας ε, τροφίμων επιδέχεται βελτιώσεις βέβαια. Αλλά μην δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα με την ασφάλεια τροφίμων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το είπε και η Κάτι άλλο σημαντικό είναι οι κυρώσει. Οι κυρώσει κάθε φορά που υπάρχουν απάτες στον τομέα των τροφίμων. Οι υπεύθυνοι πρέπει να διώκονται με υψηλές κυρώσεις, πρόστιμα κλπ. Πολύ ψηλά για να είναι και αποτελεσματικά. Τώρα πέρα από αυτά τα θετικά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που δεν βλέπω εγώ στο σχέδιο αυτό έκθεσης. Πρώτον, η θεμελιώδη συζήτηση για την διατροφική μας αλυσίδα. Και έτσι κατά πρώτον σκέφτομαι την πρόθεση μιας πιο σύντομης, πιο μικρής Αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται βιολογικά είτε οτιδήποτε άλλο, όπου να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, εφόσον ακριβώς η αλυσίδα αυτή είναι πιο κοντή. Εδώ στην Φλάνδρα υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία μας και εκείνες ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να επιβαρύνουμε αυτού του είδους επιχειρήσεις με υπερβολικές διοικητικέ διαδικασίες. Αυτό που θέλω ο καταναλωτής είναι ποιότητα. Δεν πρέπει να γίνουμε τα θύματα των απατών που κάνουν ορισμένοι. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις ετικέτες, δεν πρέπει να βάζουμε υπερβολικό άχθος στους παραγωγούς, κυρίως εκείνους οι οποίοι πάντα συμπεριφέρονται καλά. Μην ξεχνάμε λοιπόν τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να μην τους επιβάλλουμε υπερβολικό φόρτο. Ευχαριστώ. Τώρα κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η κυρία Αντελάνγκε έχει ετοιμάσει μια εξαίρετη έκθεση. Όντως και εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένας ορισμός, ένας ε, ενιαίος ορισμός. Ο κανονισμός 188-2000 λέει ότι δεν πρέπει να παραπλανώνται μέσω ε, της ετικέτας οι καταναλωτές. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τι είναι η απάτη και αφού υπάρχει και το κάτω αλιμετάριος πρέπει να διακρίνουμε την απάτη η οποία οφείλεται σε σκοπιμότητα για οικονομικό κέρδος και την απάτη η οποία δεν καταστρέφει την υγεία. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα παράπτωμα και θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Τώρα πολύ καλά τα είπε η συγγήτρια. Υπάρχει οικονομικό κέρδος στην πραγματική απάτη γιατί παραπλανάται ο καταναλωτής με λάθος ετικέτες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι εύκολα. Γίνονται απάτες στο κρέας λόγου, στο μέλι που πουλάνε κάτι που δεν είναι μελί ή στο ελαιόλαδο όπου η ετικέτα μπορεί να λέει ελαιόλαδο αλλά στην πραγματικότητα να μπερδεύεται εκεί το παρθένο ελαιόλαδο με το πυρηνέλαιο. Η απάτη είναι δύσκολο να αποφευθεί πλήρως, αλλά πρέπει να διώκεται με ελέγχου και με κυρώσεις που να είναι αρκετά αυστηρές για να είναι αποτρεπτικές για αυτόν που θέλει να εξαπατήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένα, μια μικρή παρατήρηση έχω να κάνω στην κυρία Ντελάνκε στο σημείο 27 που μιλάει για τις έρευνες και και αναφέρεται κάποια στιγμή στο Πανεπιστήμιο που το γνωρίζει καλά πολλά πανεπιστήμια και πολλά ερευνητικά κέντρα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν να μην αναφέρουμε μόνο το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και του Φάχενίγεν, αλλά να λέμε γενικά για άλλα πανεπιστήμια γιατί είναι και άλλα. Η κυρία Τεστόρντορ, η Γενική Διευθύντρια, όταν ήρθε εδώ με την κρίση του λογίσου κρέατος μας είπε ότι με την ετικέτα στην προέλευση δεν θα είχαμε αποφύγει αυτή την απάτη. Εγώ θα ήθελα να το σχολιάσει αυτό η συγκεντρία. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο και δεν θα αποφύγει την απάτη. Κυρίως για τρόφιμα, τα οποία αποτελούν σύνθεση διαφορετικών συστατικών. Η Επιτροπή τώρα θα έχει το λόγο και μετά η συγκεντρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αρχίσω πρώτα απ' όλα με ευχαριστίες προς την εισηγήτρια την κυρία Ντελάνγκε. Χαιρόμαστε που συμμερίζετε τις ανησυχίες μας όσον αφορά τις απάτες στα τρόφιμα. Είναι σαφές το ότι οι απάτες αυτές είναι επικίνδυνο και για την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και για το εμπόριο. Είναι σαφές αυτό. Επίσης Ξέρουμε ότι σε περιπτώσεις απάτης στα τρόφιμα τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα. Όμως τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι πάντα επαρκή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η επιβολή και η συνεργασία αποτελεί στοιχείο κλειδί για την καταπολέμηση των απατών αυτών. Θέλω να αναφέρω λοιπόν μερικά στοιχεία της δράσης μας. Πρώτα απ' όλα είπατε ότι πρέπει να έχουμε καλά καταρτισμένο προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Θα το συζητήσετε και σύντομα. Έχουμε την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού για τους ελέγχους που μιλάει για την παρετέρω ανάπτυξη της δυνατότητάς μας επιβολής του νόμου. Συμφωνούμε για τις κυρώσεις, συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι αποτρεπτικές και αυτή είναι και η αρχή η οποία προτείνουμε εμείς στο νέο κείμενο του νέου κανονισμού για τους ελέγχους. Επειδή 9 χρόνια όμως ήμουν επιθεωρητής στα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, πρέπει να σας πω ότι καμία κύρωση δεν αποτρέπει τους πραγματικούς εγκληματίες, γιατί θεωρούν ότι δεν θα πιαστούν ποτέ. Είναι αποτρεπτικό για αυτούς οι οποίοι σκέφτονται να το δοκιμάσουν οι άλλοι όμως, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς ε, εδώ και καιρό είναι μέσα στο έγκλημα, εκεί χρειάζονται πραγματικά καλές πληροφορίες πληροφοριών και καλή έλεγχη. Δημιουργήθηκε όντως μια ειδική μονάδα στις υπηρεσίες μας μετά την ε, απάτη με το κρέας αλόγου για να μπορούν να γίνονται ε, καλύτεροι έλεγχοι στα κράτη-μέλη και να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει βέβαια η υπόθεση αυτή να λαμβάνει υπόψη όλους τους κανόνες που ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα πολύ απλό, πάντως το δουλεύουμε. Επίσης, αρχίζουμε να φροντίζουμε και για την συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών που εμπλέκονται στο θέμα επιβολής του νόμου. Πιστεύω ότι και αυτό είναι στοιχείο κλειδί. Θέλουμε επίσης να κάνουν περισσότερες προσπάθειες στο δίκτυο ελέγχου των τροφίμων όπου συμμετέχουν οι υπηρεσίες επιθεώρησης από πλευρά των χωρών μελών. Αλλά θέλουμε συνεργασία και με την αστυνομία, τα τελωνία και άλλες ειδικευμένε μονάδες που πρέπει να ενθαρρύνουμε να συνεργάζονται όλο και περισσότερο με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τροφίμων. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι για όλα αυτά τα θέματα και για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα σε λεπτομέρειες οργανώνουμε μία διάσκεψη στη... το δεύτερο εξάμενο του 2014 υπό Ιταλικής Προεδρίας για την ασφάλεια των τροφίμων και εκεί θέλουμε να έχουμε πραγματογνωμοσύνη από ειδικού. Οπότε εξετάζουμε τέτοια τεχνική ε, πραγματογνωμοσύνη πώς ε, θα είναι διαθέσιμοι, να προσκαλέσουμε δηλαδή ειδικού και τα λοιπά στη διάσκεψη αυτή. Έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον εντοπισμό των απατών στη διατροφική αλυσίδα. Αναφέρατε διάφορα στοιχεία που είπατε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, αναρμονισμένος ορισμός ή να αναπτυχθεί περισσότερο η ιδέα των εργαστηρίων αναφοράς. Υπάρχει κάτι το οποίο ίσως να απληθει περισσοτερο η ιδεα των εργαστηριων αναφορας υπαρχει κατι το οποιο ισως να ξερετε ως refit όπου εκεί εξετάζουμε κατά πόσο είναι κατάλληλη νομοθεσία με τον στόχο στο τομέα των τροφίμων. Να λοιπόν μια ευκαιρία όπου μπορούμε να μιλήσουμε για τον εναρμονισμένο αυτό ορισμό της απάτης στα τρόφιμα. Να ξέρετε πάντως ότι η συζήτηση θα κρατήσει καιρό γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να εναρμονίσουμε τα όσα ισχύουν στο ποινικό δίκαιο των χωρών μελών και έχουν να κάνουν με απάτα στα τρόφιμα. Το θέμα τώρα των εργαστηρίων αναφοράς είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Είναι μια ιδέα που αξίζει να συζητηθεί παρετέρω. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας γι' αυτό και όπως είπα και στην αρχή, ευχαριστούμε για την έκθεση και είμαστε στη διάθεσή σας για παρετέρω συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τέλος, η εισηγήτρια. εντελάνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους για τα διάφορα στοιχεία τα οποία προσθέτουν. Είναι στοιχεία, πολλά από αυτά, τα οποία είναι παρόντα στην έκθεση, αλλά εντάξει, ίσως θα έπρεπε να υπογραμμιστούν περισσότερο. Για παράδειγμα, αυτά που είπε ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές, που θέλει μια τροποποίηση όσον αφορά το σύστημα συναγερμού. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς διατύπωση θέλετε, τι να προσθέσουμε. Εντάξει, αυτά που άκουσα δηλαδή από τους συναδέλφους λίγο πολύ υπάρχουν, αλλά ίσως ε, χρειάζεται μια διαφορετική... Το ηλεκτρονικό σύστημα δηλαδή που επιτρέπει την ταχύα ανταλλαγή πληροφοριών υπάρχει στην παράγραφο 29. Επί όσον αφορά το περίπλοκο της διατροφικής αλυσίδας που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι υπάρχει στην έκθεσή μου. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε και να δούμε μήπως πρέπει να χτενίσουμε λιγάκι την διατύπωση που χρησιμοποιούμε. Για τα παρασιτοκτόνα. Ε, διστάσαμε πολύ κατά πόσο θα έπρεπε ή όχι να συμπεριληφθεί εδώ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το πρόβλημα. Είναι όντω μια ξεχωριστή κατηγορία. Διαφορετική δηλαδή από τις άλλες περιπτώσεις απάτης στα τρόφιμα, αλλά καλά, ας το εξετάσουμε μήπως μπει εδώ. Το ίδιο και για τους φιλελεύθερους. Για, την, ε, για το επικριτικό βλέμμα όσον αφορά τους οικονομικούς περιορισμούς, δηλαδή τα χρήματα τα οποία τελικά δίνουν τα κράτη-μέλη για τους ελέγχους στα τρόφιμα. Όντω ο προπολογισμό μειώνεται συνεχώς και στη δικιά μου τη χώρα το ίδιο συμβαίνει. Έχουμε φτάσει νομίζω στον πάτο. Δεν μπορούμε να κόψουμε πια τίποτα άλλο. Η μεγάλη πρόκληση όσον αφορά τις υπηρεσίες ελέγχου είναι πώς με τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα, αλλά πώς με τα χρήματα που έχουμε μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά. Γι' αυτό σας έδωσα το παράδειγμα της Δανίας και της Ιταλίας που αντιμετωπίζουν ε, πιο με πνεύμα όμευση το θέμα των ελέγχων. Για το ECR και τον ε, το Horizon 2020 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, σίγουρα θα τη συμπεριλάβω και για τους λιανοπολιτές επίσης. Α, ναι. Όλοι αναφέρθηκαν στο θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών. Με την ετικέτα. Μπορεί να ενημερωθεί από την ετικέτα. Και τι πληροφορίες πρέπει να έχει η ετικέτα αυτή για να ενημερώνεται ο καταναλωτής. Για μένα, οι περισσότερες απάτες είναι είτε στην αρχή, στους αρχικούς παραγωγούς είτε στο τέλος πριν φτάσει στα χέρια του καταναλωτή. Ο καταναλωτής δηλαδή τελικά δεν παίρνει αυτό το, για το οποίο πληρώνει. Ενώ θα έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη στο τελικό προϊόν που παίρνει. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνήθως τα βάζουμε με τους ενδιάμεσους, με αυτούς που είναι στο μέσο της αλυσίδας. Οπότε εδώ συμφωνώ με τους συναδέρφους Και ναι, να συζητήσουμε αν η λύση είναι η επαναδιατύπωση της ετικέτας. Ο συναδέρφος από τους πράσινους λέει ναι προσοχή όμως μην επιβαρύνουμε υπερβολικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μελέτη αντικτύπου για να ξέρει τι σημαίνει η αλλαγή στις ετικέτες. Και στη δικιά μου την ομάδα, να ξέρετε, είναι πολλοί που το θέλουν. Ανεξάρτητα με το τι τελικά θα λέει η μελέτη αυτή αξιολόγησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ένα σωρό ε, μηνύματα που φτάνουν σχετικά με την αλλαγή στις ετικέτες. Πάντως για την απάτη θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό, δίχως άλλο. Και στην κυρία Γιούσο, ναι, φυσικά και υπάρχουν και πολλά άλλα πανεπιστήμια τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και της ασφαλειάς τους, της αυθεντικότητάς τους. Εγώ ανέφερα αυτά γιατί είναι αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή και συνδέουν τη γνώση από την γεωργία, από τη μια, και από την άλλη το θέμα της εγκληματολογίας, γιατί πρέπει να έχουμε αυτή την επιστημονική γνώση για να συνδέσουμε αυτά τα δύο, την γεωργική παραγωγή, αν γίνεται με το σωστό τρόπο, όπως πρέπει, και να είναι σωστό όταν λένε ότι είναι βιολογικά, για παράδειγμα, αν έχουμε και την ε, γνώση μέσω της εγκληματολογίας να είμαστε σε θέση να προσέξουμε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν απάτες για να προλαμβάνουμε τις απάτες αυτές. Γι' αυτό εγώ λέω να βγάζουμε εκτός παιχνιδιού αυτούς που έχουν την πρόθεση να εγκληματίσουν με απάτες στη διατροφική αλυσίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Στερντελάνγκε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 18 Οκτωβρίου. Στις 27 ε, Νοεμβρίου θα το συζητήσουμε ξανά εδώ και θα το ψηφίσουμε και δεν ξέρουμε πότε θα περάσει από την Ολομέλη. Και τώρα συνεχίζουμε με την ημερήσια μας διάταξη και την ΕΦΣΑ. σε σχέση με τον προτινόμενο μηχανισμό διαβούλευσης πριν από την υποβολή αίτησης για το ισχυρισμούς υγείας. Ζητήθηκε από τους συναδέλφους λοιπόν να γίνει η συζήτηση αυτή και γι' αυτό θα ζητήσω ε, από τους συναδέλφους έψα να έρθουν εδώ ή αλλιώς ε, καθίστηκε εκεί που είστε, δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ούρλα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, την ΕΦΣΑ. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ίσως η Επιτροπή και η συγήτρια της προηγούμενης έκθεσης να συγγήσουν. Ωραία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε που καλέσατε την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, για να ε, εκθέσουμε τις απόψεις μας και να σας μιλήσουμε και για τις δικές σας ανησυχίες σε σχέση με τη λειτουργία του όλου συστήματος ασφάλειας τροφίμων. Σύμφωνα με τον κανονισμό του 2006, το πεδίο εφαρμογής σχετίζεται με την ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και στα πλαίσια αυτά η ΕΦΣΑ το 2008 έλαβε 4.600 αιτήσει αξιώσεων δηλαδή και 10.000 μεμονωμένες προσφυγές πολύ περισσότερο από το προσδοκόμενο, γιατί περιμέναμε περίπου χίλιες προσφυγές. Μέσα στα τέσσερα επόμενα χρόνια, σε σχέση με, τις, ε, με τα αιτήματα υγείας, έχουμε ε, εκπληρώσει με τις υποχρεώσεις μας ε, ως προς 2.800 προσφύγες. Ως προς τον τομέα της βοτανολογικής, αυτή τη στιγμή υπάρχει στασιμότητα. Είχαμε σωρία ε, προσφυγών να αντιμετωπίσουμε, αλλά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα και το άρθρο 13.1 έχει ολοκληρωθεί με βάση τις επιστημονικές μελέτες που ζητήθηκαν. Ως προς τις προσφυγές με βάση το άρθρο 13,5 και το άρθρο 14 που σχετίζεται με την μείωση των κινδύνων ασθένειας, έχουμε λάβει ε, πολλές αιτήσει 417 προσφυγές έχουμε και έχουμε καλύψει το 40% με βάση την διαδικασία των προσφευγόντων και την αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ζήτησε και άλλο περιθώριο, δηλαδή πέντε μήνες από την λήψη των προσφυγών μέχρι του φτάσει σε συμπεράσματα και όταν ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες τότε πρέπει να σταματήσει η προθεσμία ή να δοθεί δίμηνη παράτηση. Για τους προσφεύγοντες αυτό έχει επιπτώσεις διότι οι προσφεύγοντες έχουν 15 μέρες για να υποβάλουν περαιτέρω στοιχεία. Θεωρήθηκε ε, μια επιταχυμένη διαδικασία, αλλά οι 15 ημέρες είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα και για τους προσφεύγοντες. Ως προς τις ε, προβιωτικές ε, προσφυγές, μπορούμε να πούμε ότι τα επιστημονικά κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια που ισχύουν σε ολόκληρο το νομέα υγείας. Δηλαδή, στις προσφυγές προβιωτικής ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Η ΕΕΦΣΑ έχει αξιολογήσει 300 προσφυγές προβιωτικής για, για 200 μικροοργανισμούς. Άρα το μέχρι τώρα πρόβλημα με τις προσφυγές προβιωτικής σχετιζόταν με το ότι δεν είχαμε σωστή χαρακτηριολογία των στελεχών αυτών ως προς τα προβιωτικά προϊόντα δηλαδή. Δεν είχαμε πλήρη ανάλυση των στελεχών. Έγιναν και νέες προσφυγές για επαναξιολόγηση, αλλά η έκβαση ήταν αρνητική για αυτές τις ε, προσφυγές προβιωτικής. Άρα, από πλευράς ΕΦΣΑ το σύστημα λειτουργεί καλώς. Αυτό προβλέπεται και από τις νομικές διατάξεις, το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το σύνολο των επιστημονικών στοιχείων, σταθμίζουμε δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία όπως προβλέπει ο οικονομισμός και πρέπει να γίνει η αξιολόγηση στο ανώτατο ε, δυνατό ποιοτικό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει εναρμονισμένη αξιολόγηση αυτών των προσφυγών. Και η αξιολόγηση γίνεται και προθείται στην ΕΦΣΑ και όχι στις εθνικές αρχές. Επί της ουσίας από πλευράς ΕΦΣΑ η Ευρώπη έχει προβεί σε μία συγκριτική αξιολόγηση και πολύ ζηλεύουν το ευρωπαϊκό σύστημα, άλλες χώρες και άλλες ήπειροι. Γιατί οι προδιαγραφές μας στον τομέα της υγείας είναι πολύ υψηλές και έτσι επιτρέπουμε την σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την πλήρη προστασία των καταναλωτών. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ε, είναι υπερήφανες για τα αποτελέσματα που επιτύχαμε σε σχέση με τις προσφυγές ε, στον τομέα υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ούρλ, η Επιτροπή έχει το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα υπενθυμίζω το άρθρο 6, παράγραφο 23 του κανονισμού, όπου αναφέρεται ότι οι προσφυγές θα πρέπει να αιτιολογούνται με πλήρη επιστημονικά στοιχεία και αξιολόγηση στο, σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι δραστηριότητες της ΕΦΣΑ καλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές και αυτή την εντολή και συμβαδίζουν με αυτό τον κανόνα. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η εργασία αυτή, μάλλον ο όγκος εργασίας δεν προβλεπόταν να είναι τόσο υψηλός και συμφωνούμε με τη δήλωση της ΕΦΣΑ ότι οι δραστηριότητες στέφτηκαν από επιτυχία και ότι ο κανονισμός λειτουργεί πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία ε, Αγιούζο, Τζούλι Γκέρλινγκ στη συνέχεια. Η κυρία Αγιούζο έχει το λόγο, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο και διευθυντή της ΕΦΣΑ και την Επιτροπή που προσήλθε εδώ σήμερα. Είμαι πεπισμένη ότι η εργασία της ΕΦΣΑ είναι πολύ καλή, βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και είναι, ε, διέπεται μάλλον από πλήρη διαφάνεια. Η του επίπεδου αυτή η εργασία ακολουθεί επιστημονικά κριτήρια, προβάλλει σεμινάρια και συνεδριάσεις για να πληρούνται αυτά τα κριτήρια και απαντά σε όλες ε, τις ε, προσφυγές ως προς τα προβιωτικά προϊόντα. Και όπως είπαμε και στους συντονιστές, εδώ έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Είχαμε σωρία προσφυγών και ισχυρισμών και καμία δεν εγκρίθηκε. Όμως, υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρά τα επιστημονικά στοιχεία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Ελβετία προβλήθηκε ένας ισχυρισμός επί του θέματος σε σχέση με την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμως να πω ότι μετά τις διαβουλεύσεις της ΕΦΣΑ ως προς τα επιστημονικά κριτήρια για τις ε, δηλώσεις ως προς τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τα ε, προβιατικά, θεωρούμε ότι, τα ότι αυτές οι ουσίες, τα προβιωτικά, χρησιμοποιούνται γενικά έτσι ώστε να μην γίνεται χρήση αντιβιωτικών που σχετίζονται με την ε, διάρρεια, που μπορούν να προκαλέσουν διάρρεια. Τι έγινε με αυτές τις ε, αιτήσει, τις ε, προσφυγές. Νομίζω ότι δεν ορίσαμε σωστά και δεν ξέρουμε ποια χρήση στελεχών έγινε. Γι' αυτό νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει διαβούλευση πριν από την υποβολή υποψηφιατήτων και θα βοηθήσει τους υποψηφίους να επιλύσουν μία σειρά προβλημάτων χωρίς, πριν λάβουν μάλλον αρνητική απάντηση από την ΕΦΣΑ γιατί πολλοί ιατροί και επιστήμονες και όπως είπε και η Επιτροπή Φαρμάκων υπάρχει αιτιώδη συνάφεια με την χρήση ορισμένων ε, ε, στελεχών ε, λακτόζης που ορίζονται ως προβιωτικά προϊόντα και δεν φτάσαμε σε κανένα συμπέρασμα ως προς αυτά. Μια και είναι εδώ η Επίτροπη, θα ήθελα να πω ότι μόλις ε, δημοσίευσε τον κανονισμό 907 που θα τεθεί ενισχύ αυτή τη βδομάδα σε σχέση με τη χρήση προβιωτικών και την ε, χρήση των ε, γενετικών καταστροφέων δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γενώσιμα προϊόντα σε σχέση με τα προβιωτικά. Μιλάμε για τρόφιμα ή ποτά σε ζύμωση. Τη στιγμή που γίνεται ε, ζύμωση, γαλακτοζύμωση, θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορούμε να μιλήσουμε αυτό το γενικό όρο. Θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος και ελπίζω ότι σιγά σιγά αυτά τα θέματα θα επιληθούν. Όταν μιλάμε για υγειονομικούς ισχυρισμούς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι γιατί μιλάμε και να μην υπάρχει αυτό το συγκρουσιακό καθεστώς. Julie Γκέρλιν. Ευχαριστώ. Εγώ έχω διάφορες ε, ερωτήσεις για διάφορα επίπεδα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι στιγμής ε, δεν μας λένε ε, ότι η ΕΦΣΑ έκανε άσχημα τη δουλειά της και δεν μας ανησύχησαν ότι δεν προχωρούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο η νομοθεσία δεν είναι τόσο συγκεκριμένη ε, και στην πορεία χρειάστηκε να ληφθούν διάφορες αποφάσεις για την ερμηνεία της. Δεν είναι μια ξεκάθαρη υπόθεση που λέει ε, κάντε αυτό και άρα εμείς το κάνουμε. Ακόμα και ο τόνος γενικός αποδεκτές επιστημονικές αποδείξεις μπορούμε να το συζητήσουμε πολλές ώρες. Γιατί αυτό που μπορεί εγώ να δέχομαι ή το κράτος μέλος μου μπορεί να μην το δέχεται άλλος. Και ανέκαθεν ε, ξέραμε ότι αυτό είναι δύσκολο. Νομίζω ότι και το, τα υψηλότερα δυνατά στάνταρ, οι προδιαγραφές, και αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ε, είναι θέμα προστασίας ε, καταναλωτή και δεν θέλω να φανταστεί κανείς ότι προσπαθώ να ξεφύγω από το καθήκον μου. Όχι, εγώ θέλω να προστατευτούν οι καταναλωτές. Αλλά κάποια αποτελέσματα των όσων έχουμε κάνει είναι παράξενα και προσωπικά πιστεύω πως η απόρριψη κάθε ε, ισχυρισμού περί ε, προβιωτικού προϊόντος ε, να απορρίπτεται αυτόματα ε, είναι εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά έχω πάρει τέτοια ιατρική συμβουλή από ένας από τους καλύτερους γαστρεντερολόγους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, μου είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιώ τέτοια προϊόντα. Λοιπόν, δεν λέω πως απολύτως είναι λάθος, αλλά πάντως σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο με τον οποίο τα ερμηνεύουμε εμείς όλα αυτά και με το πώς λειτουργούμε. Προσπαθώντας λοιπόν να δω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, νομίζω πως τελικά υπάρχει πρόβλημα σε διάφορους τομείς. Και το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό και η Εύσα το είχε δεχτεί, αναγνωρίσει, Στην αρχή τον ισχυρισμό υπήρχε πρόβλημα με τον όγκο, με το κατά πόσο μπορεί να κάνει να αντιδράσει γρήγορα. Υπήρχε ένα ε, πρόβλημα λοιπόν καταγραφής και, για και αυτό δημιούργησε δυσκολίες. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση της προϋποβολής το τμήμα της διαδικασίας. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πολλοί ετώντες θα προχωρούσαν στα τυφλά μέχρι στιγμής. Ε, Ένα παράδειγμα είναι η βρώμη. Η βρώμη μειώνει το κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις. Απορρίπτεται, γιατί δεν υπήρχε η άμεση συσχέτιση. Και επίσης η βρώμη μειώνει την χολυστερίνη ε, και μετά ε, μειώνει τις καρδιακές παθήσεις. Αυτό έγινε δεκτό, επειδή υπήρχε εκείνο με τη χολυστερίνη στη μέση. Αν λοιπόν από την αρχή ξέραμε πώς να τα πούμε και πώς να τα γράψουμε, ε, θα ήταν καλύτερο. Βέβαια λένε διάφοροι ότι η προϋποβολή είναι ακριβή, ότι δίνει λάθος παραπλανή ας πούμε, τον κόσμο ότι θα πάρουν την έγκριση κτλ. Πάντως ε, υπάρχουν ε, τρόποι για την προϋποβολή στα website των αντίστοιχων οργανισμών της Υπάρχει τέτοια διαδικασία και δεν βλέπω λόγο γιατί να μην μπορεί και η ΕΦΣΑ να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη διαδικασία. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή και να μας πει η ΕΦΣΑ αν πιστεύει πως κάτι τέτοιο θα βοηθήσει. Επίσης θέλω να πω κάτι ακόμα για τα υψηλ, τις υψηλότερες δυνατές ε, προδιαγραφές. Εντάξει, φυσικά θέλουμε τις υψηλότερες δυνατές ε, προδιαγραφές για τους καταναλωτές μας, αλλά υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για το ποια είναι, σε ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές. Μία είναι οι δοκιμές ελέγχου. Είναι σωστές, ας πούμε, για τη γλυκόζη, για προϊόντα όπως η γλυκόζη γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε με έναν πληθυσμό που παίρνει αυτό το υποκατάστατο για να, ε, για να είναι καλά. Και είναι κάτι πολύ διαφορετικό από όταν έχεις να κάνεις με ένα γιατρικό, ένα φάρμακο που το δίνει σε πολύ κόσμο και μετά ελέγχεις την αποτελεσματικότητα του φάρμακου πάνω στον κόσμο που έχει υποφέρει από μια συγκεκριμένη ασθένεια. Πολύ διαφορετικό πράγμα. Εάν ακολουθήσουμε αυτό το ελέγχους δοκιμίε, ε, ακολουθούμε λάθος δράμο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο χωρίς να αρχίσουμε να κάνουμε μαζικές αλλαγές στον κανονισμό. Κανένα δεν θέλει να ανοίξει αυτό το κούδι της Πανδώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα. Ανέφερα την γλυκόζη, γιατί και πάλι είναι κάτι το οποίο δεν έχει την έγκριση, αλλά εκατομμύρια καταναλωτές Ευρωπαίοι το χρησιμοποιούν. Και νομίζω πως είναι ε, ένα ωφέλιμο προϊόν για πολύ κόσμο. Και επίσης τα προβιωτικά προϊόντα εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει όφελος, δεν είναι όφελος το οποίο έχει αποδειχθεί μέσω διαδικασιών που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε, αλλά και δεν προσπαθώ να παρακάμψω οτιδήποτε ή να πω ότι ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στα προβιωτικά προϊόντα ε, υπάρχουν αποδείξεις, απλώς δεν είναι τις κατάλληλες και δεν έχουν γίνει με την κατάλληλη διαδικασία τη έρευνε Αυτά, ευχαριστώ. Η Dagmar του Parent. Ωραία, λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Ε, η Εύσα είναι παλιά ιστορία. Και μ' άρεσε που άκουσα από κάποιον που δεν είναι στην Εύσα από την αρχή ότι είναι πολύ περήφανος για τη δουλειά του. Λίγο μεγαλύτερη μετριοπάθεια δεν θα σας έκανε κακό, κατά τη γνώμη μου. Όταν ξεκινήσαμε την νομοθεσία για την ΕΦΣΑ, μπορώ να πω ότι δεν ήταν καθόλου επιτυχής η διαδικασία και καθόλου περήφανος δεν θα έπρεπε να είστε για την αρχή. Εκτός που αναγνωρίζω ότι η δομή στην ΕΦΣΑ άλλαξε όχι εύκολα, όχι εύκολα, ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πιέσουμε για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη επιστημονική ποιότητα, για ένα σωρό πράγματα. Τίποτα δεν πέρασε εύκολα. Και εκτιμώ, και λυπούμε που το λέω, πως ο διευθυντής δεν είναι πια στη θέση του, που δεν είναι πια στη θέση του, έκανε πολλή δουλειά, ακόμα και αν παρακολούθησε τη δουλειά της με συμπάθεια μένα, αλλά επιφυλακτικά. Και θα πρέπει να έρθω στη σημερινή διάταξη και να πω... Να πω και προς τη συνάδελφο Αγιούζο ότι αυτή εδώ η έκθεση δεν μιλάει για τα προβιοτικά προϊόντα, ούτε για τη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς μέσα στα προβιωτικά προϊόντα. Αν η Κομισιόν δεν μπορεί να απαντήσει σήμερα εδώ λοιπόν, την καταλαβαίνω. Στην ατζέντα αυτό έχουμε. Μιλάμε για την προϋποβολή και διαβούλευση. Θέλω να πάρω το παράδειγμα των προβιωτικών που πρότεινε η κυρία, Πρέταξη, η κυρία Γκέρλινγκ και η κυρία Γιούζο. Εγώ είμαι δικηγόρος. Κανείς μας εδώ δεν είναι επιστήμονας που να είναι σε θέση να αποφασίσει αν η ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που λέει ότι καμία από τις 300 αιτήσει που έλαβε η ΕΦΣΑ δεν, είναι, δεν έγινε δεκτή σωστά ή όχι. Κανένα από τα προϊόντα αυτά δεν θεωρήθηκε προβιωτικό και επαρκώς. Πώς γίνεται να πείτε ότι δεν, είναι, ότι δεν φέρει τα επαρκή χαρακτηριστικά. Και εδώ να σας δώσω διάφορες συμβουλές και βοήθεια. Δεν θέλω να τα πω αμέσως ότι σας κριτικάρω. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν καμιά από αυτές τις, αιτιολογι... Ε, αιτήσει είναι αιτιολογημένη ή όχι. Δεν το γνωρίζω. Αλλά εάν πιστεύετε πως οι, τα προϊόντα αυτά δεν έφεραν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, γιατί δεν το είπατε στους ετούντους και ακριβώς γιατί δεν κάνατε αυτό που σας είπαμε, δηλαδή μια διαβούλευση πριν την υποβολή. Όταν θα γίνει αυτή η συζήτηση ping-pong, γιατί φαντάζομαι πως θα μου απαντήσετε και φαντάζομαι τι θα μου απαντήσετε, θα μου πείτε ναι, αλλά η ΕΜΑ και η ΕΚΑ είναι πλούσιες υπηρεσίες γιατί ε, παίρνουν λεφτά. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι εξή, γιατί εσείς αντιπροσωπεύετε τον ε, Διευθυντή και δεν είναι και μυστικό ότι μπορεί και εσείς να θελήσετε να τον αντικαταστήσετε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, ε, δεν έχουμε χρόνο για αυτά, ας είμαστε ευθύ. Εσείς θα ζητήσετε ε, τέλη. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος που η ΕΦΣΑ δεν πληρώνεται τίποτα. Θεωρώ πως είναι λάθος μέγα. Εγώ είμαι η τελευταία που θα πω πως η υπηρεσία είναι πολύ κοντά στη βιομηχανία. Έτσι κι αλλιώ είστε κοντά στη βιομηχανία καθημερινά. Και γιατί θα πρέπει διαφορετικά από την αίμα ή την ΕΚΑ να σας ε, συγκρίνουμε. Θα ζητήσετε λοιπόν από την Κομισιόν και πάλι να εξετάσει το θέμα των τελών. Έγινε μια μελέτη αξιολόγηση, αλλά ήταν ψηλοανόητη. Ξέρω ποιος δεν ήταν υπέρ των τελών στην Κομισιόν και πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν ήμουν άμεσα πεπισμένη, αλλά μετά είδα ότι στην πράξη ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν ε, τέλη. Να σας πω κάτι ειλικρινά. Ε, εγώ είπα όχι γιατί δεν είχα εμπιστοσύνη στην ΕΦΣΑ, δεν ήξερα τι θα κάνουν τα λεφτά. Και τότε εκείνοι οι πρώτοι υπάλληλοι ήταν στο δικό τους κόσμο ήταν στο δικό τους κόσμο, δεν είχαν επαφή με την πραγματικότητα. Ελπίζω να έχει αλλάξει αυτό τώρα. Τι θα τα κάνετε λοιπόν τα λεφτά, αν πούμε ότι έχετε χρήματα. Θα δουλέψετε για τους ετούντες, γιατί αυτό παίρνε, κάνετε. Θα παίρνετε τα τέλη από τους ετούντες. Αυτό κάνει η ΕΜΑ και η ΕΚΑ και γι' αυτό και έχουν και διαβούλευση πριν την υποβολή και γι' αυτό πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να γίνεται κάτι, θα έπρεπε να είναι μια υπηρεσία την οποία προσφέρεται φυσιολογικά και πρέπει να προσέχω γιατί η Κατρίν ε, είναι πολύ υπεύθυνη. Είναι πολύ περήφανη για το γραφείο εξυπηρέτηση που έχει φτιάξει. Να υπάρχει κάποιο που να λέει: Ναι, θα πρέπει να κάνει το τάδε, να κάνει την τάδε έτσι εκεί, πόσε μέρε έχει, ποιον πρέπει να δει και σε ποιον πρέπει να μιλήσει. Εντάξει, όλα αυτά βοηθούν. Αλλά δεν είναι επιστημονικοί σύμβουλη. Αυτοί οι κακομέρδε εκεί, 6-7 πόσοι είναι, πώ θα το κάνουν αυτό στην ουσία είναι γραμματοκιβώτια. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται κάτι που θα δίνει συμβουλές στη φάση πριν την υποβολή της αίτησης. Εάν σας είχαν πει, ας πούμε, σε μια διαβούλευση πριν την υποβολή, meeting, διαβούλευση, ό,τι θέλετε, πείτε το. Έρχονται, ας πούμε, από, τους, από τα προβιωτικά προϊόντα. Α, έχετε αυτό το συγκεκριμένο ε, συνδυασμό εδώ. Ναι, το ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε την α, β, γ, δ μελέτη, για να είμαστε βέβαιοι ότι αποδεικνύεται. Πώς θα το κάνουν, πώς θα το ξέρουν, να μυρίσουν τα νύχια τους. Γι' αυτό ακριβώς λέμε για προϋποβολή. Η συζήτηση ανάμεσα σε εσά την ΕΦΣΑ και τους ετούντες, πώς να το πω τώρα διπλωματικά, ε, δεν, δεν, δεν, δεν ήταν αποτελεσματική. Ότι όλοι αυτοί οι ετούντες δηλαδή σας ενοχλούσαν. Ναι, ναι, δώστε μας την αίτηση, αλλά μην μας ενοχλείτε, θα σας καλέσουμε εμείς. Και εγώ το είδα αυτό προσωπικά. Και δεν ήταν μόνο το η αίσθησή μου, ήταν αυτό που λέγατε κιόλα, ε, γιατί το άκουσα με τα αυτιά μου. Μη μας τηλεφωνάτε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Το άκουσα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει από πλευρά ΕΦΣΑ. Εγώ πιστεύω προϋποβολή για όλα, όχι μόνο για τα προβιωτικά προϊόντα, για όλους όσους είναι οι πελάτες σας. Κάθε ετών είναι υπάλληλό σα. Η φάση της προϋποβολής είναι ουσιώδης. Μη μου πείτε δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε αυτό. Εγώ προσωπικά θα πίστευα, αν κοιτούσα το σχέδιό σας, και το οργανόγραμμά σας ότι θα μπορούσα να βοηθήσω για να το αντιμετωπίσετε, για να το καλύψετε. Δεν πιστεύω πως είστε στην ίδια κατάσταση όπως στην αρχή όταν ξεκίνησε η νομοθεσία. Σίγουρα ο κόσμος σας δουλεύει, αλλά είμαι βέβαιος πως θα μπορούσατε να, να κάνετε και κάτι παραπάνω. Η αίμα, ας πούμε, κάνει τη φαρμακοεπαγρύπνηση χωρίς να πάρει ούτε ένα τσακιστό παραπάνω για να το κάνει αυτό να το κάνετε και να πείτε μετά στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο, μα εμείς θέλουμε να, έχουμε, ε, να πληρωνόμαστε για όλα αυτά. Και μάλιστα σας συμβουλεύω να το κάνετε αυτό και γρήγορα. Και ξέρω ότι ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής μας ε, αρχίζει να ανυπομονεί, γιατί πάντα μιλάω πάρα πολύ, αλλά πραγματικά θα αντισταθώ στο πειρασμό να πω κάτι για τα τρόφιμα που είναι θρεπτικά, τα συμπληρώματα τροφών, διατροφής που συνήθως ε, ε, θεραπεύουν κάποιες ασθένειες ή καλύπτουν κάποια κενά. Και δεν αναφέρομαι καθόλου στα διάφορα βότανα και τέτοια, γιατί εκεί θα χαθούμε και η άποψή μου δεν θα βοηθήσει. <laughs> Ξεφυσάει ο Πρόεδρος. Okay, ε, jetzt möchte ich einmal EFSA. Καλώς. Να στραφώ και πάλι στην Εύσα. Παρακαλώ. Για να απαντήσετε στις διάφορες ερωτήσεις, τα σχόλια, τις ιδέες που ακούστηκαν. Παρακαλώ και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος βασικά της συζήτησης, στον τομέα δηλαδή της προϋποβολής για μας δεν είναι πρόβλημα. Προσπαθώ να καλύψω αυτά που θέσατε γενικότερα και αν χρειαστεί και ειδικότερα μετά. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι με στόχο την καινοτομία στην Ευρώπη και προκειμένου να βοηθήσουμε τους ετούντες που είναι οι πελάτες μας, συμφωνώ μαζί σας, ε, θέλουμε και πρέπει να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο αρχικό στάδιο των αιτήσεων. Δεν είναι αλήθεια ότι η δεν έχει κάνει τίποτα. Και δεν είναι όπως το λέτε κυρία Μπέρντ, ότι είναι θέμα διοικητικής βοήθειας. Όχι, είχαμε επαφές μαζί τους, όπως ξέρετε στην ιστοσελίδα μας έχουμε και διάφορα και έχουμε απαντήσει πολλές φορές στις ερωτήσεις των ετούντων. Έχουμε και workshop και μαζί τους και για μελέτες. Η ΕΦΣΑ δηλαδή έχει ήδη αναλάβει αρκετά βήματα προκειμένου να βοηθήσει τους ετούντες να καταλάβουν το σύστημα και να κάνουν ακόμα καλύτερες αιτήσει. Κάτι το οποίο είναι και προς όφελος της ΕΦΣΑ, γιατί αν έχετε μόνο καλές αιτήσει, τότε είναι προτιμότερο και για μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα σημαντικό θέμα είναι το εξή. Θέλουμε με κάθε επιχείρηση για συγκεκριμένες αιτήσει να έχουμε επαφές. Εδώ βλέπω ένα πρόβλημα. Γιατί για μένα υπάρχει και νομικό ζήτημα γι' αυτό το τέτα τέτ. Η αίμα έχει συγκεκριμένη εντολή στον κανονισμό της να έχει ένα σύστημα για εκ των προτέρων επιστημονικές συμβουλές. Δεν είναι το θέμα μόνο της αμοιβή, είναι θέμα νομικού πλαισίου. Η αίμα μπορεί βάσει του κανονισμού της όσον αφορά την καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα πριν την υποβολή να δώσει συμβουλές και έχει και το προσωπικό για να το κάνει. Εμείς στο δικό μας ιδρυτικό κανονισμό δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Τώρα υπάρχει και ένας κίνδυνος, γιατί αν έχουμε έτσι τέτα ε, με τις επιχειρήσεις πριν υποβάλουν την αίτηση και το ρώτησε και η κυρία Γκέρλινγκ εδώ βλέπω πρόβλημα γιατί νομίζω ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής δηλαδή τα μέλη του, των πάνελ δεν μπορούν να δώσουν τέτοιες συμβουλές. Εγώ δεν το βλέπω. Γιατί τα μέλη του πάνελ πρέπει να εκπονήσουν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητοι. Και ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι η ΕΦΣΑ κατά το παρελθόν χρειάστηκε να κάνει πολλά για να φτάσει στην ανεξαρτησία έκανε πολλά για να βελτιώσει την κατάσταση. Οπότε αν τώρα μπούμε σε αυτά τα τέτα τέτ, και τις συμβουλές με την ε, επιστημονική γνωμοδότηση τα μπερδέψουμε, αυτό είναι ένα θέμα. Και το τρίτο μου ζήτημα είναι το θέμα των πόρων. Αναφερθήκατε κι εσείς. Υπήρξε μελέτη αξιολόγησης τα τελευταία χρόνια και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο δυνατότητας να ζητήσουμε αμοιβή. Ίσως στο μέλλον είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως προς το παρόν δεν έχουμε. για πόσο ξέρουμε. Φυσικά και είναι θέμα πόρων. Γιατί αν είχαμε 300 ε, συναντήσεις το χρόνο, γιατί να περιοριστούμε σε έναν τομέα μόνο. Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό εγκάρσια. Και αν έχουμε συναντήσεις εκατοντάδες το χρόνο, φυσικά και υπάρχει επίπτωση στον προπολογισμό και με τον προπολογισμό που έχουμε τώρα δεν βλέπουμε να είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Συνεπώς πρέπει να βρούμε άλλα μέσα να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Να βελτιώσουμε δηλαδή την επικοινωνία, τη στήριξη στους ετούντες για όλους τους κλάδους που υποβάλλουν αιτήσει για άδειε ή για συμβουλευτικέ γνωμοδοτήσεις από την ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ να μπούμε στη συζήτηση, ευχαρίστως να κάνουμε περισσότερα, αλλά όπως είπα διστάζω να το κάνω αυτό τέτα τέτ με τι επιχειρήσει. Νομίζω ότι λείπει το νομικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και μετά ξεχνάμε ότι περνάει η ώρα και έχουμε και άλλα θέματα. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ακούσαμε πριν. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του τρέχοντος νομικού πλαισίου και των υπαρχόντων ανθρωπίνων πόρων θέλει να προσπαθήσει να υπάρχουν περισσότερες συμβουλές και περισσότερη ενημέρωση προς τους ετούντες στο σάδιο πριν από την υποβολή των αιτήσεών τους. Πρέπει να ξέρετε ότι έμαθα πως πολλά από τα θέματα τα οποία τίθεται θα μπορούσαν όντως να είχαν λυθεί πριν την... Ε, που λέμε ότι θα μπορούσαν να είχαν λυθεί στο προηγούμενο στάδιο. Δεν γίνεται γιατί ο εντοπισμός του προβλήματος γίνεται αφού έχει υποβληθεί η αίτηση. Τώρα για το θέμα της αμοιβή δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ξέρετε ποια είναι η θέση της Επιτροπής και δεν έχει αλλάξει. Ένα μόνο θέλω να πω, ότι δεν είναι μόνο θέμα εσόδων, είναι και θέμα θα βελτιωθεί η δυνατότητα ανταπόκρισης της ΕΦΣΑ. Αν κατάλαβα καλά τώρα με ρωτήσατε για γενική περιγραφή δεν έχει να κάνει με τους ισχυρισμούς για την υγεία. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο βάσει κριτηρίων που θα αξιολογηθούν από τις χώρες μέλη και όχι από την ΕΦΣΑ. Η απάντησή μου λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε μερικές περιπτώσεις να λυθούν κάποια προβλήματα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια γενική λύση για τα προβλήματα που συζητάμε σήμερα και είναι πολύ δύσκολο απριόρι να προκαταλάβω τα αποτελέσματα. Μέχρι εδώ μπορώ να πάω, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Αλλά επανέρχομαι λίγο στην γενική προσέγγιση όσον αφορά το προκαταρτικό στάδιο πριν την υποβολή αιτήσεων. Ξέρουμε ότι οι μερικές φορές διαμαρτύνονται ότι ακόμα και αν έχουν τις πληροφορίες είναι τόσο περίπλοκες που τίθεται θέμα ερμηνείας τους και κατανόησής τους. Οπότε, ίσως χρειάζεται συνεργασία με την ΕΦΣΑ για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πάντως το θέμα των ατομικών διαβουλεύσεων εξαρτάται από την ε, άποψη που έχει ΕΦΣΑ γι' αυτό. Πρόεδρος. Καλώς. Τάγμα Ροντμπέργκ πάλι. Πολύ χαίρομαι τις συναντήσεις αυτές με την Επιτροπή που τέρπουν. Δίνουν λίγο φως στις μαύρες μου μέρες. Δεν θέλω εσάς να φέρω σε δύσκολη θέση να σας βασανίσω, αλλά τους ανώτερούς σας. Δηλαδή, σε σχέση με την αυτονομία της ΕΦΣΑ που τίθεται να αμφιβόλω αν μπουν τέλη. Αλλά αυτό δεν ισχύει με, την με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή την ΕΚΑ. Γιατί πρόκειται για παρόμοιες περιπτώσεις. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ξέρουμε γιατί η μελέτη αντικτύπου ήταν αρνητική για τα τέλη που θα έπρεπε να επιβληθούν. Δηλαδή, μην το φωνάζουμε με ντουντούκα, αλλά στο λέμε μεταξύ μας. Ίσως να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στην εργασία της ΕΦΣΑ. Και αν η Επιτροπή δεν είναι έτοιμη να δει αυτό το θέμα, ε, εμείς σαν Κοινοβούλιο είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να το δούμε και η κυρία Γκέρλινγκ θα ασχοληθούν με το θέμα, καθώς και η κυρία Αγιούσο. Γιατί δεν βλέπω το λόγο, γιατί έχουμε τρεις οργανισμούς με πελάτες από τη βιομηχανία, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Βεβαίως με την φαρμακοεπαγρύπνηση υπάρχει ένα θέμα με τα χημικά και με την ΕΦΣΑ. Αλλά αυτό είναι μέρος της εργασίας. Είμαστε σε επαφή με τη βιομηχανία και θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός προπιστοποίησης ή προαδειοδότησης. Και θα ήταν πιο ειλικρινές εάν η Επιτροπή γνωρίζει ότι αυτή η διάκριση δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά από κανέναν. και μιλάτε για το ότι αντιτάσσεστε στα τέλη. Εγώ δεν λέω ότι η βιομηχανία πρέπει να καταβάλει το κόστος πάντα. Αλλά το σκέλος του πελάτη είναι σημαντικό. Η ΕΦΣΑ άλλαξε, οι πελάτες είναι περισσότεροι, είναι ένας καλύτερος οργανισμός από ότι 3, 5, 7 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ξέρετε ότι είμαι αθυρόστομη και πάντα εκφράζω την άποψή μου. Δημοσία. Εκτιμώ την εργασία της ΕΦΣΑ, μπορεί να βελτιωθεί, αλλά οι απαντήσεις σας στην ιστοσελίδα, τα σεμινάρια και ούτω καθεξής δεν με εντυπωσιάζουν. Όταν μιλάτε για μεμονωμένες ε, συναντήσεις που σας φέρνουν σε δύσκολη θέση, Μα πρέπει να δείτε και μεμονωμένες προσφυγές και αιτήσει. Δεν κοιτάτε συλλογικές μόνο αιτήσει 50 ανθρώπων, αλλά και αιτήσει του ενός. Πρέπει να μιλήσετε και με τα μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Όταν αποφασίστηκε ο οργανισμός αυτός, ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε νοσοκομείο το 2000 και όλα έγιναν πολύ καλά από τον εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ. Όμως κάναμε ένα λάθος, γιατί είναι ο μόνος ο οργανισμός ο οποίος ρυθμίζει μία αγορά όπου δεν υπάρχει προέγκριση από το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι λάθος και το έλεγα εξ αρχής. και δεν μπορούμε να, μην έχουμε σαφείς επιλογές για το τι πρέπει να κάνει η ΕΦΣΑ. Τότε ήταν ένας νέος οργανισμός. Αλλά ε, οι κανονισμοί μπορούν να αναδιατυπωθούν. Θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανονισμούς. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται. Μιλήσατε για τον κανονισμό της αίμα του Οργανισμού Φαρμάκων. Εγώ προέρχομαι από την Αυστρία και με τη Γερμανία ακολουθούμε το νόμο. Αλλά επειδή δεν υπάρχει στον κανονισμό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή μην, μην μου προβάλλετε τέτοιο επιχείρημα. Εσείς μιλάτε για το ότι δεν πρέπει να προβληθεί κάτι από το πάνελ, αλλά την αίμα τη γνωρίζω πολύ καλά. Θα μπορούσε να ισχύσει κάτι τέτοιο. Μα υπάρχει κάποιος αρμόδιος σε αυτές τις ε, συναντήσεις. Κάποιος πάντα έρχεται από την αρμόδια Επιτροπή Φαρμακευτικών Σκευασμάτων για Ανθρώπινη Χρήση. Λένε ότι η τάδε η δύναμα μελέτη δεν αρκεί ή αρκεί ως προς τη φήμη σας πρέπει να φοβόσαστε πολύ για τη φήμη σας και την ιστεροφημία σας, αλλά ε, αυτό δεν θα πρέπει να σας φοβίζει υπερβολικά. Κύριε Ούρλ, αν πούμε ότι γίνονται διαβουλεύσεις για την προπιστοποίηση, τι θα γίνει, πώς μπορούμε να περιορίσουμε. Με τα τέλη, αν θεσπίσουμε τέλη τη στιγμή που δεν υπάρχουν τέλει καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει, να το βάλουμε αυτό σε ένα αυλάκι. Αν θέλει κανείς μία διαβούλευση πριν από την υποβολή αίτησης, ποιος μπορεί να τον καθοδηγήσει με διαφάνεια. Δεν το ξέρω. Αλλά ως προς τα τέλη θεωρώ ότι πρέπει να επιβληθούν ως προς τους ε, πόρους σας, μπορείτε να ανταποκριθείτε, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε και το help desk. Δεν ξέρω κατά πόσο το χρειάζεται ε, πραγματικά και εν πάση περιπτώσει δεν θα επανεφεύρετε τον τροχό εσείς. Ε, η ΕΦΣΑ έχει το λόγο και μετά η Επιτροπή, η κυρία Γκέρλινγκ και η κυρία Αγιούσο. Ευχαριστώ. Η Ροτ Μπέρεντ έχει μεγάλη πείρα από τις απαρχές της ΕΦΣΑ. Εγώ προσήλθα σε αυτήν την επιτροπή πρόσφατα στο Κοινοβούλιο, αλλά φτάσαμε στα ίδια συμπεράσματα περίπου. Δεν είναι θέμα ιστορικού, μίσου παθών και ούτω καθεξής. Πρόκειται για μία λογική διαδικασία. Διαδικασία εκλογήκευσης. Μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας χωρίς να υπάρχει αναδιατύπωση. Θα γίνει και αναδιατύπωση, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε με μεγάλες αλλαγές. Αυτό το πνεύμα μας διέπει. Ως προς τη διαδικασία πριν από την υποβολή και κατά την υποβολή, δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ μας. Εγώ αναφέρθηκα σε έγγραφα που έλαβα από την ΕΦΣΑ πριν από 18 μήνες όταν ανέκυψε αυτό το ζήτημα. Η ΕΦΣΑ έδωσε ε, νέες σύμβουλες με βάση ένα συνεχή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, ιστότοπους, ε, απαντήσεις στην ιστοσελίδα και ούτω καθεξής. Αυτό ήθελα να εξελιχθεί για να είναι μία συνεχής φυσική εξελιχτική διαδικασία. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως προβλεπόταν. Ίσως υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι' αυτό, αλλά δεν πρέπει να διαφωνήσουμε ως προς την αρχή του να γίνει κάτι τέτοιο. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω τις εργασίες σας και θεωρώ ότι ο οργανισμός ε, τα, κατάλαβε, τα κατάφερε πολύ καλά. Και πολλοί θέλουν να μιλήσουν με τους ετούντες γιατί έτσι θα βελτιωθούν τα πάντα, τα, πάντα για τον καταναλωτή, για το κοινοβούλιο, την ΕΦΣΑ και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχετε σοβαρές αντιρρήσεις για κάτι τέτοιο. Εσείς δεν θέλετε μεμονωμένες ε, συζητήσεις με τους ετούντες, κάτι το οποίο δεν κατανοώ. Και αυτό μπορούμε να το επιλύσουμε. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχει συσταθεί η όλη διαδικασία. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσει με μονομένα φυσικά πρόσωπα. Άρα θεωρώ ότι δέχεστε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει θέληση. Μιλήσατε για μη ύπαρξη τελών. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Όλα μπορούν να αλλάξουν να υπάρχει σοβαρός λόγος. Και η εργασία της ΕΦΣΑ είναι πολυφασματική σε σχέση με άλλα ζητήματα που σας απασχολούν, όπως είπε η Πιλάρ, ας πούμε, ως προς τους ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Γιατί να μην προβάλλουμε αυτή την προσέγγιση. Άρα μπορούμε, αν το δούμε ευρύτερα το ζήτημα, να επιλύσουμε ζητήματα, γιατί στη βοτανολογία τα καταφέρατε πολύ καλύτερα. Είχαμε ένα σύστημα που θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα για να αντιμετωπίσετε με το υπάρχον σύστημα τις αιτήσει που λαμβάνετε. Ευχαριστούμε. Η Πιλάρα Γιούζο και μετά μπορεί να απαντήσει και η Επιτροπή αν το θέλει. Ευχαριστώ. Και εγώ εκτιμώ την πείρα και την παρέμβαση της κυρίας Ροντ Μπέρεντ. Εγώ γνωρίζω μόνο την ΕΦΣΑ ως οργανισμό και έμαθα πολλά, γι' αυτό ε, εκτιμώ τη δική της εργασία που έχει περισσότερη πείρα με περισσότερους οργανισμούς. Μιλήσαμε για τα προβιωτικά, γιατί το θέμα μας απασχόλησε στους συντονιστές σε σχέση με τους ισχυρισμούς που προβάλλονται για τα προβιωτικά. Συγκεκριμένα, ως προς τις πρώτερες διαπραγματεύσεις Θεωρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται αυτές οι προγενέστερες διαβουλεύσεις. Μπορούν να είναι και μεμονωμένες να αφορούν μια ομάδα επιχειρήσεων ή όχι. Συμφωνώ με τις προλαλήσασες και να καλύπτονται και τα έξοδα για αυτές τις διαβουλεύσεις, διότι η επιχείρηση ή ο τομέας θα πρέπει να πληρώνει για μια προγενέστερη διαβούλευση, διότι έτσι θα εξοικονομήσουν χρήματα μέσα στα πλαίσια της αίτησης και δεν θα γίνονται άσκοπες ε, συναντήσεις ή δωρεάν διαβουλεύσεις, οι οποίες δεν επιλύουν προβλήματα πάντα. Η ΕΦΣΑ για άλλη μια φορά, ο κύριος Ούρλ Ευχαριστώ. Εάν συνοψίσω, μπορώ να πω ότι δεν διαφέρουμε πολύ. Έχουμε τον ίδιο στόχο, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες. Όπως είπε η κυρία Γκέρλινγκ, κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και η κυρία Αγιούσο αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως δεν χρειάζεται να μιλάμε σε μεμονωμένες, με μεμονωμένες επιχειρήσεις. Ίσως μπορούμε να μιλήσουμε σε έναν όμιλο επιχειρήσεων που έχουν τις ίδιες προθέσεις. Και αυτό έχει το θετικό ότι μπορούμε να ομαδοποιήσουμε. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε σε πόρους και ως προς την αντίληψη που έχουμε. Χαίρομαι για τη συζήτηση αυτή, γιατί και εμείς ε, θέλουμε να μάθουμε από τις δικές σας προσδοκίες. Συμβαδίζουμε και όσον αφορά την Εύσα μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Κυρία Γκέρλιν, θα προσπαθήσουμε με εργαστήρια να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα ήθελα να πω όμως ότι χρειάστηκε να εργαστούμε με βάση 4.000 αιτήσει, άρα ήταν δύσκολο να γίνει ταξινόμηση Τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο να επανέλθουμε στο ζήτημα, όπως είπε και η Επιτροπή. Ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς ξαναβλέπουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για να γίνει πιο σαφές αυτό. Έτσι ώστε να δούμε τα ε, ε, θέματα που μας απασχολούν περισσότερο με σοβαρότητα Ίσως να μην είμαστε τόσο γρήγοροι, αλλά στο τέλος θα φτάσουμε στο στόχο που εκφράσατε. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank. Ähm, ich weiß es weitere Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση συμπληρωματική. Ναι, μπορώ η κυρία Ντακμαρ Μπέραντ. Μέχρι τι 18.30 έτσι καλώ έχουμε, 6.30 έχουμε την αίθουσα. Ντακμαρ Μπέραντ. Κοιτάξτε, θέλω μια διευκρίνηση. Λέτε ότι δεν θα υπάρξουν ατομικά συναντήσεις, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη συνάντηση με όλες τις επιχειρήσεις μαζί. αν μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι εντάξει κάποιου η πρόταση και σκεφτείτε ότι θέλετε να αφήσετε μόνες τους τις επιχειρήσεις, εγώ νομίζω ότι όχι, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Δεν είναι μια καλή ιδέα. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Δεν είμαι αφελής, ξέρω τι εννοείται, το καταλαβαίνω και όχι, δεν είναι αυτό που λέμε. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο στόχος μιας συνάντησης πριν υποβληθούν οι αιτήσει. είναι για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εμείς δεν θα κοιτάξουμε τις μελέτες, δεν θα τις αξιολογήσουμε, δεν θα δώσουμε ενδείξεις για το κατά πόσο θα είναι χρήσιμες ή όχι. Όχι, πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα, να πούμε τι είδους ε, μελέτες θέλουμε, πώς να είναι φτιαγμένες, τι στατιστικές θέλουμε και με τις πληροφορίες αυτές οι ετούντες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις κατάλληλες μελέτες. Προς το παρόν, όταν έχουμε προβλήματα, είναι να έχουμε μελέτες που δείχνουν τη σχέση ανάμεσα στην αιτία και το αιτιατό. Αυτά τα προβλήματα δεν τα λύνουμε όταν έχουμε ήδη τις μελέτες. Όχι, πρέπει να αρχίσουμε νωρίτερα να έχουμε επαφές με τους ανθρώπους αυτούς για να τους εξηγήσουμε πώς θα κάνουν κατάλληλες για μας μελέτες. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με περισσότερους ετούντες χρόνος η λύση δηλαδή δεν είναι μόνο το φαρμακευτικό που σκεφτόμαστε που είναι η αίμα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τρόφιμα και φάρμακα είναι διαφορετικά. Η καινοτομία είναι διαφορετική στη μία και στην άλλη περίπτωση. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να εφαρμόζουμε το ίδιο σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά με την αίμα να θέλουμε να το εφαρμόσουμε και στην ΕΦΣΑ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία για να πετύχουμε τον ίδιο στόχο. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Κύριε Ροτβέρεντ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Φτάνει. Η επόμενη συνεδρίαση 24 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ όλους σας που μείνατε εδώ μέχρι το τέλος. 21 Οκτωβρίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. 9 με 12. Όσοι θέλουν, ευχαρίστως. Έληξε συνεδρίαση, καλό βράδυ.